Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα περνάμε στις ερωταπαντήσεις. Και υπενθυμίζω στους συναδέλφους που θα λάβουν το λόγο για τις ερωτήσεις να περιορίζονται σε ερώτηση ενός λεπτού ώστε να μπορέσει να κρατήσει τα δύο λεπτά στη διάρκεια των απαντήσεων της υποψήφια. Επίτροπος, ο κύριος Βιέφκα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε υποψήφια, έχουμε νέες προτάσεις για την εταιρική διακυβέρνηση, οι οποίες θα πρέπει, πιστεύουμε, να ε, επικεντρωθούν στην ε, λειτουργία των επιχειρήσεων σε μια ενιαία αγορά, και να δώσουν περισσότερες ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανταγωνιστικότητα και ευκαιρίες μέσα σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, καθώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν τις περισσότερες εργασίες εργασία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας, θα πρέπει να αποφύγουμε την επιβολή υπερβολικών νομοθετικών ρυθμίσεων, ε, γραφειοκρατικού φόρτου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει άλλωστε και να αποδιαρθρωθεί ο εφιστάμενος γραφειοκρατικός φόρτος. Δεν ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώς μπορείτε και αν θεωρείτε ότι είναι προτεραιότητα η αποδιάρθρωση του γραφειοκρατικού φόρτου και τι μπορεί να κάνετε, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι μια υπεύθυνη προσέγγιση για τις νέες νομοθετικές προτάσεις για την εταιρική διακυβέρνηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να εκμεταλλευθώ την ευκαιρία και την χαρά να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Θα απαντήσω στα τσεχικά λοιπόν. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Σβιεύκα για την ερώτηση. Συμφωνώ πολύ για τα όσα είπατε και τις θέσεις ε, σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να φροντίζουμε όλες οι προτάσεις, οι στάση νομοθεσία να μην επιβαρύνουν περισσότερο γραφειοκρατικά αυτές ακριβώς οι επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να αποδιαρθρώσουμε αυτά τα ε, βάρη και να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ε, λειτουργήσουν και να εργαστούν πιο αποτελεσματικά μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό είναι η αρχή της περικοπής της γραφειοκρατίας και της κατάργησης αυτών των φραγμών. Έχουν ήδη κατατεθεί από την αντίστοιχη Γενική Διεύθυνση πολλές προτάσεις και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξέρουμε ότι υπάρχουν επίσης για τους αυτοαπασχολούμενους ε, συστάσεις που βρίσκονται υπό επεξεργασία. Υπάρχουν προτάσεις για τη διαδικασία της πτώχευσης για, την, ε, για διαφορετικές ρυθμίσεις στη διαδικασία της πτώχευσης και επίσης ε, διευκολύνσεις ε, οι οποίε θα έχουν να κάνουν με προβλήματα στη ρευστότητα των επιχειρήσεων, ώστε να μην αναγκάζονται να κηρύσουν πτώχευση επιχειρήσει για λόγου περιστασιακή ρευστότητα. Επίση, έχουμε να κάνουμε με τα ε, ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα των μετόχων. διαδικασίε οι οποίε θα πρέπει να απλουστευτούν πιστεύουμε. Και θέλω να επισημάνω ότι όλα αυτά πρέπει να τα υποστηρίξουμε, πρέπει να προαγάγουμε λύσεις αποτελεσματικές και πιστεύω ότι μια ε, δημόσια διοίκηση έχει σαν αυτοματισμό το να προξενεί νέο γραφειοκρατικό βάρος και εμείς πρέπει να το καταπολεμήσουμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Εύελιν Ρέγνερ από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ. Η ερώτησή μου αφορά το Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο οι εταιρείε και οι μέτοχοι ζητούν να σταθεροποιηθεί το ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο ώστε να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές περιβάλλον και να ρυθμιστούν αποτελεσματικά οι ε, σταθερά οι επιχειρηματικές του δραστηριότητε. Θα υποστήριζατε λοιπόν την ανάπτυξη περισσότερων πιο σταθερών ρυθμίσεων και ασφάλειας δικαίου για τις εταιρείε και τους μετόχους, σε παραδείγματι με τη μορφή μιας οδηγίας για τις διασυνοριακές μεταφορές εδρών εταιριών και δεύτερον μια οδηγία που να εξασφαλίζει ελάχιστες προδιαγραφές για την εμπλοκή των μετόχων και την ε, παρακολούθηση μιας προτάσεως για την ενιαία ευρωπαϊκή εταιρεία ή την ευρωπαϊκή έδρα, ώστε να μην έχουμε ζητήματα εικονικών εδρών, ε, τις λεγόμενες εταιρείες ε, ταχυδρομικό κουτί, και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι μέτοχοι θα λαμβάνουν ουσιαστικά αποφάσεις με στόχο την ε, υγεία, υγιή λειτουργία μιας εταιρείας. Πώς αλλιώς άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς όπως ο καταναλωτής, οι τοπικές κοινωνίες, οι εργαζόμενοι μπορούν να εμπλακούν στη λειτουργία μιας επιχειρήσεως. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημά σας. Συνδέεται με κάτι που είπα προηγουμένως. Νομίζω ότι οι πόροι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντικοί. Είναι 170 εκατομμύρια επιχειρηματίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ναι. Και επομένως θα πρέπει να τους δώσουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να μην αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να προτείνουμε απλοποιήσεις ιδίω για τις διαμεθοριακές αγορές οι οποίες λειτουργούν στην εσωτερική αγορά. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε την ψηφιακή αγορά. Όλα αυτά είναι δυνατότητες που έχουμε για να μπορέσουμε να άρουμε τα, τους φραγμούς που εμποδίσουν τις επιχειρήσεις να λειτουργούν σε διαμεθοριακό επίπεδο. Επιπλέον, θα πρέπει να μειωθεί η φορολογία των επιχειρήσεων. Είναι ένα από τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το δικό μου τομέα, γιατί έχω μια μεγάλη εμπειρία για την πρόσβαση στην, στα διαφθορτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την πρόταση αυτή που έχει να κάνει με τη μεταφορά των εδρών των επιχειρήσεων εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. <clears throat> Όταν μια επιχείρηση θέλει να μετακινηθεί σε ένα άλλο κράτος μέλος θα είναι υποχρεωμένη να κλείσει την επιχείρηση και να ανοίξει μια νέα επιχείρηση στο νέο κράτος μέλος. Όλα αυτά είναι θέματα που από νομοθετική άποψη θα έπρεπε να λύσουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε συνεργασία με τα κράτη-μέλη για να επιτύχουμε μια κοινή ρύθμιση για όλες αυτές τις επιχειρήσεις σε σχέση με το δικαίωμα εγκατάστασης και σε σχέση με τη λειτουργία των ε, μετόχων. Εδώ πάλι πρέπει να έχουμε νομοθετικές προτάσεις ώστε να υπάρξει σεβασμός των δικαιωμάτων των μετόχων. Ο κύριος Φως από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ. Και η δική μου ερώτηση συνδέεται με το προηγούμενο ερώτημα κυρία Γεωούροβα. Το Φεβρουάριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την άποψή του για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Αγοραστών και αυτό είχε ένα τεράστιο αποτέλεσμα ιδίως στο ηλεκτρονικό ε, ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά γενικά και στο λιανικό εμπόριο, αύξησε το διαμεθοριακό εμπόριο. Πώς λοιπόν εσείς θέλετε, βάσει και των προτεραιοτήτων της ε, Κομισιόν Juncker, να κινηθείτε για να επιταχύνετε τις διαδικασίες αυτές και να τις επηρεάσετε με θετικό τρόπο. Και ένα δεύτερο θέμα, σε σχέση με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην ισότητα των δικαιωμάτων και την, τον σεβασμό των συμβάσεων σε όποιο κράτος μέλος και αν έχουν συναυθεί. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει την απαραίτητη προτεραιότητα η σωστή εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Εσείς θα φροντίσετε για να υπάρξει η σωστή εφαρμογή και ο έλεγχος σωστής εφαρμογής στα κράτη-μέλη να ενισχυθεί αυτή η διαδικασία, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φως για το ερώτημά σας. Εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι η πρόταση σε σχέση με το δικαίωμα, με το δίκαιο των διαμεθοριακών πωλήσεων είναι πια ευρωπαϊκό δίκαιο γιατί έχει εγκριθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι δόθηκε πράσινο φως για το ζήτημα αυτό γιατί για μένα αυτό είναι ο σωστός δρόμος με τον οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε και να δώσουμε και μεγαλύτερη έμφαση στην ηλεκτρονική οικονομία, που είναι μια προτεραιότητά μας. Να απαραίτητο λοιπόν να μπορέσουμε να προωθήσουμε την πρόταση αυτή και τα κράτη-μέλη να έχουν ναι. τα κράτη-μέλη να έχουν ομοιόμορφα πρότυπα για τις πωλήσει αυτές. Για τις διαμεθοριακές πωλήσει είναι πιο εύκολο λοιπόν να το επιτύχουμε και θα είναι λιγότερο δαπανηρό για τις επιχειρήσεις και θα είναι και φυσικά και προς το όφελος των καταναλωτών. Το δίκαιο λοιπόν των πωλήσεων ήταν κάτι το οποίο επικρίθηκε από πολλούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είπε ότι δεν υπάρχει ένα εναλλακτικό σύστημα με αυτόν τον τρόπο και στράφηκαν εναντίον της ομοιογενοποίησης του δικαίου αυτού. Ενώ υπάρχει και η αντίθετη άποψη ότι πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο για την εναρμόνιση. Και φυσικά μέσα σε όλα αυτά θα πρέπει να σκεφτόμαστε πώς θα μπορέσουμε να απλοποιήσουμε τις πωλήσει μέσω διαδικτύου, το ηλεκτρονικό εμπόριο, ώστε να ενισχύσουμε αυτή την οικονομική δραστηριότητα και το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να επίσουμε τα κράτη-μέλη ώστε να δεχτούν αυτή την πρόταση η οποία μπορεί πράγματι να ενισχύσει τις οικονομίες όλων των κρατών μερών. Αν σκεφτούμε τι σημαίνει κάτι τέτοιο στην πράξη, αυτό θα δώσει δυνατότητα σε μια επιχείρηση που λειτουργεί σε διάφορα κράτη-μέλη να εφαρμόζει ένα ενιαίο δίκαιο και επομένω να δώσει στου πελάτε τη και του καταναλωτέ την ίδια πληροφορία και την ίδια ασφάλεια. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ θετικό. Uh, η κυρία Δελβό από τους Ελιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σας. Κυρία Γιώργοβα. Για τα δημόσια έγγραφα. Ξέρετε ότι σε πρώτη ακρόαση χαιρέτησε το Κοινοβούλιο την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απλούστευση και την αποδοχή ορισμένων εγγράφων στο δημόσιο χώρο και την έχει διευρύνει σε ορισμένα τη σημεία. Η απερχόμενη Επιτροπή ε, επέκτηνε την ιδέα της δημοσίευσης και το ζήτημα του κόστους της ε, ε, μετάφρασης. Εμείς θέλουμε να διευκολύνουμε λοιπόν ως προς την πρόσβαση, να διευκολύνουμε τη δουλειά των ε, επιχειρηματιών, την κινητικότητα, να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία. Τι γνώμη έχετε για αυτόν τον κανονισμό και τι είδους πρωτοβουλίες μπορούμε να εξασφαλίσουμε όσον αφορά την αναγνώριση, αμοιβαία αναγνώριση των δημοσίων εγγράφων και εάν σκοπεύετε να προωθήσετε την αναγνώριση εταιρικών σχέσεων σε μια τέτοια πρόταση. Ευχαριστώ κύριε Αντελβό. Χαίρομαι και στην υπόθεση αυτή είναι ξεκάθαρε και θετικέ οι θέσει και οι στάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. να αναγνωρίσουμε λοιπόν τι είδου αντίκτυπο μπορεί να έχει στην καθημερινή ζωή του απλού πολίτη αυτή η υπόθεση. Θα έχει τεράστιο αντίκτυπο, θα μειώσει σημαντικά την γραφειοκρατία Γιατί τώρα ξέρετε η κατάσταση είναι ότι όταν κάποιος ε, παραδείγματι ε, συνάπτει γάμο με κάποιον από διαφορετική χώρα ή θέλει να κάνει μια εταιρεία έξω από τα όρια της ε, χώρας του ή έχει ζητήματα κληρονομικού δικαίου που ξεπερνούν πάλι τα σύνορα της χώρας του, υπάρχουν πολλές περιπλοκές. Πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος λοιπόν πιο απλουστευμένος για την επικύρωση και την επικυρωμένη μετάφραση το, το, λεγόμενο αποστήλ, δηλαδή τη σφραγίδα της ε, αναγνώρισης, της αμοιβαίας αναγνώρισης των εγγράφων. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά τόσο το ιδιωτικό δίκαιο όσο και το ε, εταιρικό δίκαιο και εδώ μπορούμε να διευρύνουμε όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες το ε, φάσμα των εγγράφων που θα καλύπτονται από αυτή την αμοιβαία αναγνώριση. Ελπίζω ότι θα υιοθετήσει το Συμβούλιο τις προτάσεις αυτές. Προς το παρόν όμως ξέρετε υπάρχει η, η γνώμη που επικρατεί είναι ότι θα πρέπει να περιορίσετε μόνο στα ζητήματα του αστικού δικαίου των ιδιωτών, των ατόμων καλύτερα, δηλαδή στα οικογενειακά ζητήματα περισσότερο και όχι στα εταιρικά. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ευχαριστώ. Τρεις βασικές προτεραιότητες ε, ε, περιλαμβάνονται στην ατζέντα για τα θέματα δικαιοσύνης μέχρι το 2020. Υπάρχει το θέμα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης πάντως επί της οποίας εδράζεται η πολιτική μας στον τομέα της δικαιοσύνης οι νομικοί και οι πολίτες και οι δικαστές δεν έχουν μερικές φορές δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε άλλες χώρες. Συνεπώς απαιτούνται δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων και τη διευκόλυνση της εφαρμογής τους. Τι άποψη έχετε για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσετε να ενισχύσετε την αμοιβαία εμπιστοσύνη στις αποφάσεις των διαφόρων χωρών. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί και μέσω της ενίσχυσης των, των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας και όχι να δημιουργήσουμε νέα μέσα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν πολιτικά με στρεβλό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Λέει υποψηφία επίτροπος η ερώτηση αυτή αναφέρεται σε αυτό που είπα και πριν, δηλαδή την αναγνώριση των δημοσίων εγγράφων περισσότερο. Θα έπρεπε να συμπληρώσω αυτά που είπα και να τονίσω ότι απαιτείται πράγματι να υπάρξει αύξηση και βελτίωση των επιπέδων εμπιστοσύνης ανάμεσα στα διαφορετικά όργανα των κρατών μελών. Έχετε απολύτως δίκιο όταν λέτε ότι η αμοιβαία αναγνώριση των δημοσίων ε, αποφάσεων, των δικαστικών αποφάσεων και των δημοσίων εγγράφων ε, πρέπει ε, να γίνονται σεβαστά. Αυτό σημαίνει αμοιβαία εμπιστοσύνη, αυτό σημαίνει αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στα διαφορετικά δικαϊκά συστήματα. Εμπιστοσύνη στην ανεξαρτησία τους και στην δυνατότητά τους να εφαρμόζουν σωστά τις αποφάσεις. Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρξουν κάποια επιπλέον ε, νομοθετικά βήματα εδώ και είναι επίσης απαραίτητο να διασφαλιστεί σωστότερη εφαρμογή των νομοθετικών αποφάσεων έτσι ώστε να μην ενισχύσουμε μόνο το μέσο αλλά να ενισχύσουμε την ουσία δηλαδή την εφαρμογή της για την δημιουργία καλύτερων επιπέδων εμπιστοσύνης. Εγώ νομίζω ότι σε αυτό αναφέρθηκα στην εισαγωγική μου ομιλία. Συνεργασία, συντονισμός στα θέματα της δικαιοσύνης όπως και στα θέματα της κατάρτισης των λειτουργών της δικαιοσύνης. Ε, επίσης γενικά λίγο εδώ να τονίσω ότι ακόμα και η σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση θα βοηθήσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η επόμενη ερώτηση. Ο κύριος Κοφεράτη από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Γιούροβα. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νομοθετικής περίοδου υιοθετήσαμε διάφορα μέτρα τα οποία ενίσχυσαν το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Ανάμεσα σε αυτά είναι οι μηχανισμοί εναλλακτικών ε, επιλύσεων των διαφορών και μάλιστα για την εφαρμογή της, εφόμενης, της αυτής θα πρέπει να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η νέα. Τα νέα μέτρα αυτά όμως ίσως να μην επαρκούν να δώσουν στους ε, πολίτες τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους και στον τομέα της δικαιοσύνης και στον τομέα του κόστους της χρήσης τους. Τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε για να διαβεβαιώσετε τους Ευρωπαίους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, ότι θα έχουν τα μέσα να πρασπιστούν τα δικαιώματά τους. Οι διαδικασίες συλλογικής αποζημίωσης θα βελτιώσουν τις δυνατότητες των πολιτών ιδιαίτερα σε ό,τι έχει σχέση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σκοπεύετε να κάνετε κάποιες προ... προτάσεις γύρω από τον τομέα των συλλογικών αποζημιώσεων. Κυρία Γιούροβα. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προωθήσει διάφορα μέτρα προστασίας των καταναλωτών και των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της δυνατότητας πρόσβασής τους είτε σε δικαστικό επίπεδο ε, επίλυσης διαφορών είτε σε εναλλακτικό επίπεδο. Ε, σαν παράδειγμα έχουμε ξεκινήσει και με την εξέταση των θεμάτων επίλυσης διαφορών online όπως λέγαμε δικτυακά. Ιδιαίτερα για μικρές διαφορές, ε, κάτι το οποίο θα επιτρέψει στους καταναλωτές χωρίς ιδιαίτερο κόστος να μπορέσουν να αποζημιωθούν από πιθανές βλάβες τις οποίες έχουν υποστεί ε, σε χαμηλό επίπεδο. Αυτό δεν θα ισχύει βέβαια για ποινικού χαρακτήρα θέματα και διαφορές. Λοιπόν τώρα για τις συλλογικές αποζημιώσεις. Έχω την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη κυκλοφορήσει μία ανακοίνωση και παρακολουθεί ε, στα διάφορα κράτη-μέλη τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα των συλλογικών αποζημιώσεων είναι ένα μέσο το οποίο θα μπορούσε να συνδράμει τους καταναλωτές έτσι ώστε να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους με συλλογικό δηλαδή ισχυρότερο συνεπώς τρόπο. Εξετάζουμε λοιπόν την εφαρμογή αυτής της δυνατότητας και θα δούμε αν κάτι τέτοιο είναι χρήσιμο και υπάρχει η βούληση θα βελτιώσουμε με συμπληρωματικές προτάσεις την κατάσταση. Το θέμα είναι να έχουμε εγγυήσει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια τέτοια μέθοδος με αποτελεσματικό τρόπο. Ε, Ευχαριστώ. Κυρία. Κυρία υποψήφια επίτροπε. Είπατε ότι αν εγκριθεί η υποψηφιότητά σας το σχέδιο δράσης για, την, ε, για το εταιρικό δίκαιο θα συνεχιστεί. Περιλαμβάνει και την ε, κωδικοποίηση του εταιρικού δικαίου. Είναι αυτό μία από τις προτεραιότητές σας και εάν ναι, τι, πού θα βρίσκεται το πλεονέκτημα για την, μέσα από την κωδικοποίηση του δικαίου για τις εταιρείες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα δεύτερο στοιχείο, όλες οι επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχυθούν, να επεκταθούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν να αντιμετωπίσουν λοιπόν οι ρυθμιστικές προκλήσεις και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την άποψή σας, τι θα πρέπει να γίνει για να εξασφαλίσετε ότι θα υπάρξει μια σύγκληση σε παγκόσμιο επίπεδο των ρυθμίσεων για το δίκαιο των επιχειρήσεων μαζί με τους εταίρους μας. Και αυτό θα ευνοήσει τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτουργούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Έχω πράγματι έχω ήδη απαντήσει για τις προτεραιότητες που έχω διατυπώσει. Ο στόχος μου είναι να εξασφαλίσω την μέγιστη δυνατή προσέγγιση και σύγκληση μεταξύ τους των νομικών συστημάτων και του εταιρικού δικαίου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είπα αυτό γιατί είναι σαφές ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την ενιαία εσωτερική αγορά και η εσωτερική αυτή αγορά θα πρέπει να είναι πραγματικά μια αγορά χωρίς φραγμούς. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τις ε, συνθήκες για την λειτουργία των επιχειρήσεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μίλησα για κωδικοποίηση του δικαίου στον εμπορικό τομέα, αυτό το οποίο εγώ είχα στο μυαλό μου ήταν το στόχο που θα πρέπει να θεσπίσουμε και να θέσουμε στον εαυτό μας. Βέβαια, προτού να υπάρξει κάποια εναρμόνιση, κάποια προσέγγιση σε ό,τι αφορά τα εθνικά δίκαια, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να το συζητήσουμε αυτό και μέσα και με τα κρατημέλη, ώστε να γίνει αυτή η προσέγγιση με τον κατάλληλο τρόπο. Δηλαδή να απλοποιήσουμε τα πράγματα για τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι που θα πρέπει να πετύχουμε. Αυτό είναι ο στόχος μας. Φυσικά υπάρχει πολλής δρόμος να διατρέξουμε ώστε πράγματι να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα καταλήξουν σε αυτό το κοινό στόχο. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν σε ποιο βαθμό μπορούμε να έχουμε αυτό το κοινό εταιρικό δίκαιο που θα δώσει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις τώρα και την ανταγωνιστικότητά τους έναντι άλλων επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι δεν φέρουν πρόσθετο άχθος οι επιχειρήσεις σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχουμε τονίσει αυτό και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι για τις δραστηριότητες εξαγωγικού χαρακτήρα στην παγκόσμια αγορά δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε πρόσθετο βάρος που θα τις εμποδίσει. Από την ομάδα των ε, Φιλελευθέρων, κυρία Βίξτρομ. Thank you very much and thank you. Here I am. Straight ahead. Here I am. Good to see you and thank you for... Σας ευχαριστώ. Με βλέπετε. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είχατε το θάρρος να είστε και επαγγελματικοί σε αυτά που είπατε αλλά και προσωπικοί μέσω των περιπέτειών που μας εκθέσατε των προσωπικών σας. Υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης των εθνικών δικαστικών συστημάτων. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της ε, αμοιβαία ε, χρήσης των βέλτιστων πρακτικών. Αυτό θα βοηθήσει την εξέλιξη και την ε, ανάπτυξη μάλλον της εσωτερικής αγοράς και θα βελτιώσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και έναν πίνακα επιδόσεων στον τομέα της δικαιοσύνης σχετικά με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είστε σαν επίτροπος λοιπόν υπέρ του να συνεχίσουμε ε, την βελτίωση του ε, πίνακα αυτού επιδόσεων. Ναι, ευχαριστώ κυρία Βέικστρομ, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Σχετικά με τον πίνακα επιδόσεων, νομίζω ότι αυτό το Justice Scoreboard είναι πράγματι ένα μέσο για να αξιολογήσουμε σωστά ε, την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των εθνικών συστημάτων. Είναι κάτι που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται τα συστήματα δικαιοσύνης και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, κάτι το οποίο δεν αναφέραμε ακόμα. Ε, έχει σημασία λοιπόν αυτός ο πίνακας ε, καταγραφής των επιδόσεων. Τώρα το πώς θα συνεχίσουμε τη χρήση αυτού του μέσου στο μέλλον. Η αίσθησή μου είναι ότι παράλληλα με αυτό υπάρχουν και διαφορετικά μέσα για να βεβαιωθούμε για την σωστή χρήση ε, των κανόνων που έχουν σαν στόχο τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνουμε, ε, μια προσπάθεια που θα πρέπει να κάνουμε με τη συνδρομή των ίδιων των κρατών μελών για το αν θα πρέπει να διευρυνθεί ε, το πίνακας αυτός συμπεριλαμβάνοντας και διαφορετικούς τομείς όπως το ποινικό δίκαιο, ε, το ποινικό κομμάτι. Νομίζω ότι πράγματι αυτό θα ήταν θετικό, θα πρέπει να συλλέγουμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα, και άλλα στοιχεία, άλλα δεδομένα, άλλα στατιστικές για να αξιολογήσουμε την κατάσταση στα κράτη-μέλη χωρίς ε, ε, να προχωρήσουμε στην ε, λήψη συμπληρωματικών μέσων. Ευχαριστώ. Επέμονος ο μιλητής είναι ο κύριος Μαστάλκα εκ μέρους της ομάδας της ΓΚΟΕ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και καλή μέρα κυρία Γιώργοβα. Στις γραπτές απαντήσεις, μεταξύ άλλων, προβαίνεται σε μία δήλωση για το πρόγραμμα REFIT, ένα μέσο της εκ των υστέρων αξιολόγησης των, του αντικτύπου υφισταμένων διατάξεων. Η αποδιάρθρωση του γραφειοκρατικού φόρτου, η απλούστευση γενικά των διοικητικών διαδικασιών μπορεί να συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες. Πώς όμως μπορείτε να βελτιώσετε τις προδιαγραφές στις σχετικές με τα δικαιώματα των εργαζομένων, φερρυπίν, υγεία και ασφάλεια, κοινωνικός διάλογος. Απάντηση. Για το πρόγραμμα REFIT πρώτα. Το οποίο αποτελεί πιστεύω ένα σημαντικό μέσον για να απαντήσουμε στο ερώτημα εάν ένα σχέδιο νομοθεσίας ή ε, ε, ή προτινόμενες νέες διατάξεις εξυπηρετούν τον στόχο για τον οποίο σχεδιάζονται. Αυτό είναι ένα από τα κύρια μελήματα της Επιτροπής Juncker. Θα αξιολογήσουμε δηλαδή την ε, σκοπιμότητα, τη χρησιμότητα των νέων διατάξεων και σε αυτό θα συνεργάζομαι εκ του σύνεγγης με τον ε, Αντιπρόεδρο Τίμερμανς με τον οποίο έχουμε ήδη συζητήσει διεξοδικά το θέμα. Τώρα το πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ε, ε, τήρηση των δικαιωμάτων, το σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την, το ότι δεν θα υποβαθμιστούν οι συνθήκες εργασίας και ασφάλειας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να αντιμετωπίσουμε. και θα το πράξουμε στηριζόμενοι και στην υποστήριξη, στην αρρωγή των τομεακών οργανώσεων και ενώσεων που ε, αγωνίζονται για τα δικαιώματα των εργαζομένων και βέβαια και των συνδικαλιστικών σωματείων. Έχω πολύ καλές επαφές ήδη ακούσει από διάφορες οργανώσεις και με μεγάλη προσοχή πάντοτε ακούω τις συστάσεις εκείνων με τους οποίους ε, πρόκειται να συνεργαστώ. Επομένως, είτε πρόκειται για μη κυβερνητικές οργανώσεις, είτε πρόκειται για συνδικάτα, θα είναι πάντα χρήσιμη και κρίσιμη η συμβολή τους. Για τους εργοδότες τώρα. και τους μετόχους δεν πρέπει ποτέ να μειώνεται η πρόσταση. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ερώτηση είναι από την κυρία Χάουταλα των Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή ασχολείται όλο και περισσότερο με ε, συμβάσεις, συνθήκες περί με διάφορες χώρες. Αυτές οι ρήτρε ε, διαιτησίας που προβλέπονται σε τέτοιου είδους συνθήκες, ε, για σας τι αξία έχουν, πώς τις βλέπετε και τι σχέση έχουν με τα ένομα συστήματα των κρατών και ο πρόεδρος Γιούνκερ ξέρουμε ότι έχει εκφράσει μια δυσφορία στο να στηρίζεται ένα σύστημα σε ε, ιδιωτικού είδους δικαστήρια, τα οποία δεν καλούνται καν να αιτιολογήσουν τις αποφάσεις τους. Θεωρείτε λοιπόν ότι θα μπορούσε το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο να ενισχύσει την ευρωπαϊκή διάσταση των εθνικών μας δικαστηρίων ώστε να στηρίζονται σε αυτά περισσότερο επιχειρήσεις και όχι σε κάποια ιδιωτικά δικαστήρια σε ένα σύστημα διαιτησίας. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Το αναφέρατε και εσείς στην ερώτησή σας. Είναι σαφές από την ε, πολιτική τοποθέτηση του Ζων Κλωτιούν και ότι θα χρειαστεί για την προσεχή επιτροπή να προβλέπονται οι ίδιες οι δυνατότητες για τους πάντες. Δυνατότητες για την επίλυση διαφορών, είτε πρόκειται για εταιρείε ε, μικρές ή μεγάλες, χωρίς φραγμούς. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω τόσο, είπε ο Πρόεδρος Γιούνκερ. θα πρέπει να αποφύγουμε η αδίποτε ε, καταστρατήγηση της νομοθεσίας ή ε, οποιοδήποτε σύστημα το οποίο θα αντιπαρερχόταν τα δικαστηριά μας. Η διαιτησία είναι φυσικά ένα πολύ καλό σύστημα για την επίλυση των διαφορών, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί ως η μόνη δυνατότητα για τους εμπλεκόμενους, για τα εμπλεκόμενα μέρη. Είναι σαφές αυτό και από τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε αυτό δεν ξέρω αν μπορεί ο κανονισμό Βρυξέλλε 1 να αποτελέσει επαρκέ μέσο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων επίλυση διαφορών, που είναι το κύριο μέσο που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την ε, επίλυση διαφορών μεταξύ δύο μπλεκομένων μερών αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να ισχύσει για, δια, για ε, υπερσυνοριακές διαφορές. Κυρία Φεράρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εσείς θεωρείτε ότι η διαφάνεια και η ανεξαρτησία είναι θα έλεγα βασικά θέματα και αυτό το εκτιμάμε. Από ό,τι φαίνεται όμως εσείς για να υπερασπιστείτε τον αρχηγό του, κόμματό, του κόμματός σας, τον κύριο Μπάμπης, ήσασταν υπεύθυνοι και για την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού. Είχατε πει ότι είχε πουλήσει τις ε, επιχειρήσεις του, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε ότι οι δραστηριότητες αυτές δεν είχαν ε, ε, δοθεί, αλλά σύν της άλλης έπαιρναν χρήματα και από κοινοτικά όργανα. Πώς μπορούμε εμείς να πιστεύουμε τις μελλοντικές σας διαβεβαιώσεις. Madam, you have Ευχαριστώ. Πρέπει να είναι σαφές σε όλους. Ο Αντρέι Μπάμπης είναι ο πρόεδρος της πολιτικής κίνησης του πολιτικού κόμματος με το οποίο εγώ συνδέομαι τα τελευταία χρόνια και είμαι αντιπρόεδρος αυτού του κινήματος. Και θα παραιτηθώ βέβαια από αυτό το αξίωμα τις επόμενες μέρες. Ήταν ένα άτομο που είχε μεγάλη επιτυχία στον κόσμο των επιχειρήσεων και εμένα δεν με ενδιέφερε το θέμα των επιχειρησεών του. Με ενδιαφέρει ο πολιτικός του, το πολιτικό του έργο. Είναι υπουργό προπολογισμού στην ε, χώρα μου και αρχηγός αυτού του κόμματος. Το αν έχει πουλήσει ή όχι αυτές οι επιχειρήσεις, αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να το επιλύσει όταν ανέλαβε το έργο του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Και οι πληροφορίες που έχω είναι οι καλύτερες πληροφορίες που μπορώ να έχω για το θέμα αυτό μετά από τη συζήτηση που έγινε στο Τσεχικό Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά. Μερικές φορές γίνεται μια συζήτηση η οποία περιστρέφεται γύρω από το αν είμαι ή δεν είμαι η, αν θέλετε, η υπαρχηγός του κυρίου Μπάμπης. Όχι, εγώ σας λέω ότι είμαι ένα ανεξάρτητο άτομο και ποτέ δεν έχω υποχωρήσει ενώπιον οποιασδήποτε πίεσης ούτε του κυρίου Μπάμπη ούτε κάποιου άλλου. Και φυσικά και στο έργο μου ως υπουργό δεν έχω επηρεαστεί από κανένα και δεν ε, έχω κάποιο άλλο στόχο από το να ενισχύσω την ανεξαρτησία μου. Και σας λέω ότι τέτοιου είδους πιέσεις τις έχω υποστεί και στο παρελθόν και έχω αποκτήσει μια κάποια ανοσία σε αυτές. Αυτή τη στιγμή όμως σας λέω αυτό το οποίο εγώ γνωρίζω. Και εγώ δεν έχω ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις του κύριου Μπάμπης. Ο κύριος Βιεύκα από το ΕΛΚ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Γιαόροβα, ένα ερώτημα το οποίο συνδέεται με αυτό το οποίο είπατε μόλις. Της γνώσης σας για το ευρωπαϊκό δίκαιο. Λέτε ότι το δικαίωμα αυτό είναι αποτελεσματικό όταν μπορούν τα άτομα πράγματι μπορεί να προσφύγουν βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου όταν χρησιμοποιείται. Αλλά έχουμε κάποια εργαλεία, κάποια πιο πολύπλοκα από τα άλλα όπως η Βρυξέλλες 1 ή ο κανονισμός για τις διαμεθοριακές υποθέσεις και εδώ το ερώτημα μου είναι το εξής <clears throat> σε γενικές γραμμές. Εσείς θέλετε να θεσπίσετε κάποιες κατευθύνσεις για τους πολίτες ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν θετικά τα εργαλεία αυτά και να έχουν ε, ικανοποιητικά αποτελέσματα για αυτούς. Μα γιατί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δημιούργησαν αυτά τα εργαλεία αν δεν είναι αυτός ο στόχος τους. Ευχαριστώ λέει κυρία Γεώροβα. Κύριε Ζιεύκα, Πράγματι, ο νόμος είναι αποτελεσματικός μόνο εφόσον εφαρμόζεται και υπάρχει έλεγχος εφαρμογής του. Αν υπάρχει καθυστέρηση στην εφαρμογή του νόμου, υπάρχει ουσιαστικά απουσία της νομοθεσίας. Είναι σαν να μην υπάρχει νομοθεσία. Πρέπει να εφαρμόζεται με ταχύτητα και αυτό ισχύει και για το, τις Βρυξέλλες 1 και άλλα νομοθετικά μέτρα όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινή ζωή των πολιτών μας πρέπει να υπόκεινται σε αυτή την προϋπόθεση της ταχείας εφαρμογής. Σε αυτό το τομέα λοιπόν θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλα αυτά τα μέτρα, όλες αυτές οι διατάξεις και οι πρόνοιες εφαρμόζονται με αποτελεσματικό τρόπο. Γιατί αφορούν όλους τους πολίτες μας και θα πρέπει να έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για την εφαρμογή τους. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών μας για τις περιπτώσεις που υπάρχει κάποια αστοχία του αστικού δικαίου. Το δίκαιο θα πρέπει να αντανακλά τις ανάγκες των ανθρώπων στην, πρακτή, στην πρακτική τους καθημερινότητα. Όταν εγκρίνουμε διατάξει του αστικού δικαίου οι οποίες είναι αναποτελεσματικές στην πράξη, θα πρέπει οι πολίτες να μας το επισημαίνουν. Συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια πολύ αποτελεσματική εκστρατεία. Θα πρέπει να αυξήσουμε τη συνειδητοποίηση μεταξύ των πολιτών μας για όλα αυτά τα θέματα και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και οι νομομαθείς και οι εργαζόμενοι στον τομέα του δικαίου έχουν την κατάλληλη κατάρτιση για τα θέματα αυτά και επειδή εγώ έχω ε, σπουδάσει νομικά και ήμουνα νομομαθής στο παρελθόν, θα εξασφαλίσω ότι πράγματι έτσι είναι. Περνάω τώρα την Προεδρία και το σφυράκι στον αγαπητό μου συνάδελφο Κλοτ Μωράες, τον πρόεδρο της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Θεμάτων. Thank Σας ε, ευχαριστώ. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας καλωσορίσω και εγώ κυρία Γιάουροβα εξ ονόματος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ δικαιοσύνης και δημοσίων ελευθεριών. Τα θέματα της δικαιοσύνης φυσικά είναι κομβικά για μας. Είχαμε ήδη κάποια ανταλλαγή απόψεων και κατανοείται ότι βρίσκονται στο κέντρο της συνεργασίας μας. Η δικαστική συνεργασία στα αστικά και στα ποινικά, τα θεμελιώδη δικαιώματα και νέοι δυναμικοί τομείς όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων σε δικτυακό επίπεδο είναι βασική στόχοι για μας και είναι τα θέματα τα οποία μας έχουν ήδη και σας έχουν απασχολήσει από ό,τι φαίνεται από αυτά τα οποία είπατε. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν, ο κύριος Άξελ Φως. Ευχαριστώ. Και αφού λόγω χρόνου δεν μπόρεσε να απαντηθεί η δεύτερη μου ερώτηση, θα την επαναλάβω. Σκοπεύετε να ασχοληθείτε με τον έλεγχο και την επιβολή της ε, Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στα κράτη-μέλη. Είναι πάρα πολύ σημαντική για μένα η ερώτηση. Έχω και άλλες ερωτήσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μάρτιο ε, ψήφισε μια έκθεση για την υπόθεση NSA και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, προωθήσει το θέμα και να καταθέσει το ταχύτερο δυνατό νέες προτάσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων με βάση τις αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου και ένα επίπεδο ε, αξιόλογο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όταν θα έχετε λοιπόν την συζήτηση για τη συμφωνία σε κοινέ προδιαγραφές θα προωθήσετε την έκθεση αυτή και επίση σκοπεύει να κάνει, θα σκοπεύετε ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνετε μια νομοθετική πρόταση ώστε μέσα από ένα νομοθέτημα να θεσμοθετηθούν αυτές οι αρχές. Τρίτο τμήμα της ερώτησης, το τμήμα της προστασίας των καταναλωτών επηρεάζονται οι προσφορές προς καταναλωτές με διαφημιστικούς ε, τρόπους που έχουν να κάνουν και με τα συστήματα αναζήτησης στο διαδίκτυο ε, και θα ήθελα να σας ρωτήσω στο πεδίο αυτό πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Απάντηση. Ναι, εάν αντελήφθην σωστά έχετε διατυπώσει τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη είχε να κάνει με το πώς θα χειριστώ το θέμα της υλοποίησης της επιβολή του ευρωπαϊκού δικαίου. Βεβαίως και θα το πράξω. Υπάρχουν χρήσιμα εργαλεία σε επίπεδο ευρωπαϊκής, στη διάθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η φάση της υλοποίησης μπορεί να μην είναι μια ε, φάση η οποία έχει πολύ μεγάλη ε, επικοινωνιακή αξία ή δεν προβάλλεται ιδιαίτερα, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη ουσιαστική σημασία. Η ιδέα του ασφαλούς ε, λιμένος επίσης είναι ένα από τα πιο περίπλοκα ζητήματα, ένα από τα θέματα όπου η προστασία των προσωπικών δεδομένων και του ιδιωτικού βίου των συμπολιτών μας ε, διακυβεύεται. Εδώ πρόκειται για ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα που αναγνωρίζει ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. ώστε να υπάρχει ασφάλεια ε, για το τι γίνεται όταν φεύγουν τα δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και πρέπει να δούμε αν είναι ασφαλής αυτός ο ασφαλής λιμήν. Βλέπω από πολλούς από σας ότι υπάρχουν ε, σοβαρές επιφυλάξεις για την εφαρμογή αυτής της αρχής. Έχω και εγώ σοβαρές επιφυλάξεις. Δεν μπορώ να σας πω σήμερα ότι θα πρέπει να καταργηθεί η αρχή του ασφαλούς λιμένα ή η νομοθεσία σχετική. Όχι. Αλλά ας αναλυθεί πρώτα σοβαρά. Και ας βρούμε πρώτα ένα άλλο καλό εναλλακτικό μέσο. Εάν λοιπόν επιβεβαιωθώ ε, με εγκρίνεται στη θέση αυτή, θα ήθελα να συνεχίσω ο διάλογο αυτών και να προχωρήσω σε μια διεξοδική ανάλυση του κατά πόσον είναι ασφαλές το σύστημα αυτό και τι άλλες λύσεις θα μπορούσαμε να βρούμε, ποια άλλη, ποιον άλλο δρόμο για να βρούμε ένα καλό και αποτελεσματικό σύστημα. Βλέπω ότι έχει τελειώσει ο χρόνος μου για τις ε, μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο όμως. Ε, ε, μακάρι να μου τη ρωτήσει κάποιος άλλος την ερώτηση γιατί είναι ένα τεράστιο ζήτημα, πολύ σημαντικό και θα ήθελα να απαντήσω πιο δεξαδικό. Ε, ξέρετε ότι μου άνοιξαν τα μάτια, μου άνοιξε τα μάτια η απάντηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε σχέση με την Google και τα προσωπικά δεδομένα, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο από ό,τι βλέπω. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριο Μωρέ. Ήταν περίπλοκο το ζήτημα, σα δείχνω μια κάποια επίκαια Από του οριστέ Δημοκράτε. η επόμενη ερώτηση από τον κύριο Κλοντ Μωρέ, τον υποφινόμενο δηλαδή. Να δούμε αν μπορώ και εγώ να ε, περιοριστώ στον χρόνο μου, μια και χτυπάω το σφυράκι στον κύριο Φω για τον ασφαλή λιμένα και το ζήτημα της ε, αποκατάστασης, δικαστικής αποκατάστασης, για να επανέλθουμε όπως φαντάζομαι θα θέλετε και εσείς στο θέμα αυτό. Ε, κάποια από τα αισθήματα που έθιξε ο κύριος Φως και οι ανησυχίε του δεν έχουν καλυφθεί ακόμη. Ε, στο ζήτημα λοιπόν της έκθεσης του με την ομπρέλα προστασίας, τον ασφαλή λιμένα, είναι ζητήματα τα οποία έχουν ανοίξει, δεν έχουν κλείσει ακόμα και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θέλουμε κατεπηγόντως να αναλυφθεί δράση και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επίτροπος που να έχει σαν ε, αντικείμενο του, χαρτοφυλακίου του, την, ε, χαρτοφυλακίου του την απευθείας επικοινωνία με το Κοινοβούλιο και τα προβλήματα που εντοπίζει το Κοινοβούλιο και το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το σύνολο των προβλημάτων που επισημαίνω εγώ στην δική μου έκθεση. Είδατε 57 δευτερόλεπτα ακριβώς. Απάντηση. Σας ευχαριστώ. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε υψηλό επίπεδο προστασία. Αυτό πρέπει να, πρέπει να προβλέπει και να διαφυλάσει και η οποιαδήποτε νέα πρόταση για την προστασία των δεδομένων. Πρόκειται για έναν τομέα που μοιράζεται στις αρμοδιότητες διαφόρων επιτρόπων και είχα επικοινωνία με τον κύριο Ανσίπ που είναι συνυποψήφιος και αυτός επίτροπος και έχουμε συμφωνήσει πως εφόσον, επιλεγούμε, εφόσον εκλεγούμε θα αναλάβουμε δράση κατά τρόπο συντονισμένο και συνεργατικό. Αμέσως μόλις αναλάβει καθήκοντα η νέα επιτροπή θα ξεκινήσουμε τη δουλειά αυτή για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως όταν αυτά ε, διασχίζουν τον Ατλαντικό. Γιατί είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, αλλά και η εμπιστοσύνη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ. Μια εμπιστοσύνη η οποία πρέπει να πω ότι έχει πληγεί αρκετά. Λόγω του σκανδάλου Σνόουντεν, και άλλων σκανδάλων που αποτελούν σαφή μηνύματα πως οι υπηρεσίες των ΗΠΑ σκοπεύουν να αξιοποιούν τέτοια δεδομένα για λόγους ασφαλείας μεν, αλλά και κατά τρόπο προληπτικό, χωρίς να γνωρίζουν ε, εξ αρχής ε, σε τι μπορεί να χρησιμεύσει το δεδομένα αυτά, θέλουν να τα συλλέγουν. Είναι πολύ περίπλοκο λοιπόν το ζήτημα που θα έχουμε να επιλύσουμε τις ΗΠΑ, αλλά σας διαβεβαιώ ότι δεν πρόκειται να προβώ σε ουδεμία παραχώρηση όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ευχαριστώ. ECR Κυρία Γιώργα πιστεύω το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης είναι ένα σημαντικό εργαλείο στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και του ε, οργανωμένου εγκλήματος. Δεν είναι τέλειο όμως αυτό το εργαλείο και αναρωτιέμαι αν η Κομισιόν θα λάβει υπόψη τις ε, ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναλογικότητα αυτού του εντάλματος, ιδίως για ίσονα εγκλήματα, αδικήματα μάλλον. Επίσης στον τομέα της δικαιοσύνης, η Κομισιόν στο παρελθόν έχει αφιερώσει σημαντικούς ε, πόρους σε ε, σχέδια που ερχόντουσαν εκ του παρελθόντος, όπως ήταν ο κοινό νόμος πολίσεων και ο Ευρωπαίος Εισαγγελία. Μήπως θεωρείτε ότι χρειάζεται να υπάρξει μια αναθεώρηση όλων αυτών και όχι να δώσετε προτεραιότητα σε προτάσεις που δεν μου φαίνεται ότι είναι σημαντικές για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε δυσκολίες στο νομικό ε, σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσω εάν εγκρίνεται την υποψηφιότητά μου. Το να δω λοιπόν αν υπάρχει πραγματικά χρησιμότητα και σωστός αντίκτυπος για όλα αυτά τα σχέδια. Για μένα αυτό είναι το ουσιαστικό σε σχέση με το ευρωπαϊκό ένταλμα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι βασικό. Και έχουμε να εξετάσουμε το κατά πόσο αυτό το ευρωπαϊκό ε, ένταλμα μπορεί να τύχει της σωστής ε, ε, εφαρμογής. Και επίσης και ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει να δούμε κατά πόσον είναι πράγματι χρήσιμος και δεν είναι απλώς σε σχέση ότι πιάνουν τόπο τα χρήματα των φορολογουμένων. Αλλά πιστεύω στο παρελθόν ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα έχει ένα ιστορικό επιτυχία. Ήταν ένα εργαλείο πάρα πολύ σημαντικό για να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα στην Ευρώπη. για να εξασφαλίσει ότι οι εγκληματίες στην Ευρώπη δεν μπορούσαν να διαφεύγουν από τη μία χώρα στην άλλη. Είναι ένα αποτελεσματικό λοιπόν εργαλείο, κατά την άποψή μου, νομίζω ότι είναι περίπου 50.000 τέτοια εντάλματα που εκδίδονται κάθε χρόνο. Σε ό,τι αφορά τώρα την αναλογικότητα της χρήσης αυτού του εντάλματος, του ευρωπαϊκού εντάλματος. Φυσικά, αν εφαρμόζεται σε θέματα που αφορούν μικροποσά ή είναι ίσονα θέματα ως αδικήματα, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε ώστε να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του εντάλματος. Για να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι θα συμβάλλει στην βελτίωση της απόδοσης δικαιοσύνης. Αυτό πρέπει να κάνουμε, ποτού κάνουμε αλλαγές όμως. Από τη φιλελεύθερη ομάδα η Σόφη Βέλτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήλθατε κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Γιούγκερ σας, μας ζήτησε να βάλουμε προτεραιότητες στα πλαίσια της οδηγίας εναντίον των διακρίσεων. Παρ' όλα αυτά η ομάδα των ενδιαφερομένων πολιτών εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα ομοφοβίας και σε επίπεδο οικογενειακού δικαίου και σε σχολεία και σε γενικότερες άλλες εκφάνσεις της κοινωνίας. Πάρα πολλοί νέοι έχουν εμπόδια να αντιμετωπίσουν όταν θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην ελευθερία και ε, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επί των συνθήκων έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις και την ομοφοβία. Έχουμε ζητήσει να υπάρξει ένα και στα πλαίσια της έκθεσης Λούνατζεκ πρόσφατα ένας οδικός χάρτης για το σερασμό των δικαιωμάτων αυτής της κατηγορίας. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Πράγματι, είπατε πολλοί πράγματα τα οποία δεν θα χρειαστεί εγώ να επαναλάβω. Η οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων είναι το βασικό μέσο το οποίο καλούμεθα να χρησιμοποιήσουμε και είναι κάτι το οποίο μπορεί να καλύψει τα κενά τα οποία υπάρχουν σήμερα. Τώρα στις ερωτήσεις σας κάπως πιο συγκεκριμένα. Αυτό δεν ήταν μια δική μου πρωτοβουλία, αλλά παρόλα αυτά ε, κατανοώ πλήρως την στρατηγική η οποία ακολουθήθηκε για την αντιμετώπιση των θεμάτων που ε, έχουν μπροστά τους αυτή η κατηγορία πολιτών από ό,τι γνωρίζω υπάρχουν ίσως και 25 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών που θα έπρεπε να έχουν απολύτως τα ίδια δικαιώματα, ισότιμα δικαιώματα και θα πρέπει να προστατεύονται από ομοφοβικές επιθέσεις. Ο οδικός χάρτης τώρα στον οποίο αναφερθήκατε είναι κάτι το οποίο εάν υπάρξει θα πρέπει να έχει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη μορφή. Όπως ε, σας είπα, ε, θα πρέπει να έχουμε κάποιες συγκεκριμένες προτεραιότητες και μία ανάλυση των ε, επιθυμητών δράσεων και ευθυνών, δηλαδή το ποιος θα είναι υπεύθυνο για συγκεκριμένες δράσεις και για την εφαρμογή της στρατηγικής. Είναι λοιπόν σαφές ότι θα πρέπει εμείς να ζητήσουμε εδώ κυρίως την συνεργασία των κρατών μελών. Και νομίζω ότι κάποιες χώρες είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν. Άλλωστε και οι χώρες μέλη είναι και υπεύθυνε για τα μέσα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση φαινομένων ομοφοβικών επιθέσεων. Ε, και πρέπει να υπάρξουν φυσικά και εκστρατείες πληροφόρησης, ενημέρωσης, δημοσιεύσεις, οδηγίες, συστάσεις. E. Ευχαριστώ για την ΚΟΕ, e, η κυρία Βεργιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για την κυρία Γιούροβα, διαρωτώ με για το περιεχόμενο του χαρτοφυλακίου σας. Δίνουμε μεγάλο βάρος στις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές, τα δικαιώματά τους, ε, το κράτος δικαίου. Ε, νομίζω μέσα από το πρίσμα αυτό είναι κάτι που μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση. Γιατί έτσι και αλλιώς το θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να συγκεντρώσει την προσοχή μας. Ένα παράδειγμα να σας φέρω μετά και από αυτά που είπε η κυρία Ιντβελτ για τους Ρωμά. Είναι ο πληθυσμός ο οποίος υφίσταται τα, τις περισσότερες διακρίσεις. Ο δικός χάρτης υπάρχει, η στρατηγική υπάρχει, οι επιμέρους στρατηγικές έχουν, ε, στατιστικές μάλλον, μας δείχνουν δραματικές καταστάσεις και για πρώτη φορά στον συγκεκριμένο τομέα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια διαδικασία επί παραβάση και αφορά τη δική σας χώρα, την Τσεχική Δημοκρατία. Αυτό είναι μια σοβαρή πρόκληση για σας. Πώς θα προχωρήσετε λοιπόν στον συγκεκριμένο τομέα, πέρα από την οδηγία που έχουμε στη διάθεσή μας, τι σκοπεύετε να κάνετε έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικά και τον Ρωμά ειδικότερα.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 Νομίζω ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός των παιδιών Ρωμά πηγαίνουν σε ειδικά σχολεία και καλούμεθα να διορθώσουμε την κατάσταση. Ε, δεν θέλω να υπερασπιστώ εγώ την τσεχική κυβέρνηση, αλλά ελπίζω να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και στα πλαίσια της δίμηνης προθεσμίας που έχει δοθεί στην τσεχική δημοκρατία να έχουμε καλά νέα. Είναι πράγματι δύσκολη η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Ρωμά. Η ξεκάθαρη στρατηγική ε, από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υιοθετηθεί και από τα κράτη-μέλη. Πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν από το ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι το εθνικό και το τοπικό. Έχω αρκετή εμπειρία εδώ γιατί έχω εργαστεί σε τοπικό επίπεδο για πάρα πολλά χρόνια αλλά ε, κάτι το οποίο ελείπει εδώ είναι η εμιβαία κατανόηση ανάμεσα στην πλειοψηφία και την μειοψηφία. Βέβαια η συζήτηση αυτή ξεπερνά το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Τζιν Λάμπερτς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ την υποψήφια για την απάντησή της που αφορά τον οδικό χάρτη για τους ομοφιλόφιλους λεσβείες παρενδυτικούς και φιλομεταβατικούς. Θα ήθελα να αναφερθώ στα θέματα της οριζόντιας οδηγίας. Είχατε δηλώσει στις γραπτές απαντήσεις ότι υπάρχουν πολιτικά, πολιτική φραγμή. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε πώς σκοπεύετε να εισαγάγετε σε νομοθετικό επίπεδο και θα ήθελα και λίγο περισσότερη διαφάνεια αν μπορείτε για το ποια είναι τα κράτη που δυσκολεύονται να δεχθούν τις προτάσεις. Ίσως χώρες οι οποίες δεν έχουν δυσκολίες να ε, μπορέσουν να εκφράσουν περισσότερη υποστήριξη προς εσάς και με την κοινωνία βέβαια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που να μπορούσατε να προχωρήσετε περισσότερο. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ποιους, σε ποιους υπολογίζετε για την αρρωγή στην προσπάθεια για την καταπολέμηση των διακρίσεων ώστε να υλοποιηθεί το γράμμα και το πνεύμα του άρθρου 2 της συνθήκης για την ισότητα. Ευχαριστώ πολύ. Η οριζόντια οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Όπως γνωρίζετε. Αντιμετώπισε αντίθεση από αρκετά κράτη-μέλη Και εδώ εγώ θέλω να προωθήσω και να ολοκληρώσω το έργο αυτό σε ένα ορατό μέλλον, μέλλον το οποίο όμως δεν μπορώ να προβλέψω αυτή τη στιγμή, αλλά έχω υπόψη μου κάποιο χρονοδιάγραμμα. Κάποια κράτη-μέλη επιβάλλουν εμπόδια. Έχουν τους λόγους τους. Και επιτρέψτε μου τώρα να σας εκθέσω και από τη δική μου προσωπική εμπειρία. Ολοκλήρωσα τις ε, σπουδές νομικής, όπως σας έλεγα, σχετικά αργά στην ε, σταδιοδρομία μου, ενώ το αρχικό μου επάγγελμα είχε να κάνει με τον πολιτισμό και την ανθρωπολογία. Μπορώ λοιπόν να σας πω ότι κάθε κοινωνία σε κάθε κράτος μέλος έχει τα ιδιαίτερά της χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τις παραδόσεις του κράτους, τις συνήθειες και τα ταμπού που υπάρχουν τα οποία όμως θα πρέπει να μπορεί κανείς να ξεπεράσει. Θα πρέπει να είμαστε σε να συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη για να δούμε τι είδους φραγμοί ή εμπόδια υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ. Σας παρακαλώ να τελείτε το χρόνο σας, κυρία υποψήφια. Και το υποψήφια το τονίζω. Η κυρία Κριστίνα Βίνμπερκ εκ μέρους των EFTD. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εφαρμογή του άρθρου 21 προς το παρόν της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια ανομαλία. Αντί να έχει κανείς το δικαίωμα να επισκέφτεται κανείς τους συγγενείς του σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διεκπαιρεώσει επιχειρήσεις ή να ταξιδέψει, ουσιαστικά έχει δοθεί το δικαίωμα εισβολή σε άλλες χώρες, εργασία στη μαύρη αγορά, εκτέλεσης εγκλημάτων ή επαιτίας. Επίσης συνδέεται με ένα θέμα το οποίο πολύ σύντομα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ξέρω ότι πολλά κράτη-μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια αυτού του έτους. Αυτό είναι ο κοινωνικός τουρισμός ή ο τουρισμός για τα κοινωνικά επιδόματα. Επειδή αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το χαρτοφυλάκιό σα, θέλω να θέσω το ερώτημα αν θα αντιμετωπίσετε τι γελίε αυτέ τι συνέπειε του άρθρου 21 κατά τη διάρκεια τη θητεία σα. Θα ήθελα εδώ να πω ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων είναι μια θεμελιώδης αρχή για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω αναλύσει την κατάσταση <clears throat> σε διάφορα κράτη-μέλη. Όταν προσπαθούσα να αναλύσω το θέμα αυτό της ελεύθερης κυκλοφορίας, αυτό το οποίο διαπίστωσα είναι ότι τα κράτη-μέλη έχουν πολύ καλά εργαλεία στην διάθεσή τους για να αντιμετωπίσουν πιθανές καταχρήσεις. Και έχουν δύο συγκεκριμένα εργαλεία στη διάθεσή τους για να αξιολογήσουν το κατά πόσο η συμπεριφορά των ανθρώπων που εισέρχονται στη χώρα τους έρχεται σε σύγκρουση με τις αρχές της ε, δημόσιας τάξης. Και επίσης <clears throat> τίθεται το ερώτημα του κατά πόσο αυτά τα άτομα καταχρώνται του συστήματος κοινωνικής προνοίας. Και εκεί πάλι τα κάτι μελέχουν τα απαραίτητα εργαλεία και θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν όταν έρχονται σε ε, αντιμετωπίσουν περιπτώσεις που είναι σαφής ε, καταχρήση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. Κάτι το οποίο έχει συμβεί σε πολλές χώρες. Πιστεύω λοιπόν ότι το θέμα αυτό απαιτεί καλύτερη παρακολούθηση. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι η Κομισιόν αξιολογεί τώρα περιπτώσεις καταχρήσεως του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας σε διάφορα κράτη-μέλη και θα καταλήξει σε μια πρόταση για να επιληθεί το πρόβλημα αυτό, χωρίς φυσικά να θίξει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας. Εάν η κατάσταση φτάσει απαράδεκτα επίπεδα και χρειάζεται μια νομοθετική πρωτοβουλία, αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να συμβεί. Σύμφωνα όμως με τις πληροφορίες μου είναι επαρκής η ισχύουσα νομοθεσία για να αντιμετωπίσει τέτοιε περιπτώσεις. Για τους μη εγγεγραμμένους, η κυρία Βίκη Μέιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως ε, Επίτροπος το θεμετοφύλαξ των συνθηκών και η ισότητα είναι πολύ σημαντική μέσα στη συνθήκη αυτή. Δέχεστε ότι το Ισλάμ δεν αναγνωρίζει την ισότητα ανδρών και γυναικών και το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι μετανάστες που έρχονται από Ισλαμικές χώρες έχουν σαν αποτέλεσμα να υποσκάψουν την ισότητα που έχουμε επιτύχει για τα θέματα αυτά. Είναι κάτι το οποίο θα είναι στο θεματολόγιο των ε, προτάσεών σας. Ε, Είμαι πεπισμένη, λέει κυρία Γιώουροβα, <clears throat> ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν την ίδια υποχρέωση να σέβονται τους νόμους και τους κανόνες που εφαρμόζονται στους ε, ηθαγενείς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν έλθουμε ενώπιον περιπτώσεων που υπάρχει παραβίαση αυτών των κανόνων, έχουμε τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις περιπτώσεις αυτές. Δεν είμαι το κατάλληλο άτομο για να αξιολογήσω την ε, φιλοσοφία του Ισλάμ και άλλων θρησκειών. Αλλά Εφόσον μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα άτομα αυτά θα πρέπει να σέβονται τους ίδιους κανόνες όπως και οι άλλοι πολίτες ανεξάρτητα της θρησκευτική τους πίστης. Τα δικαιώματα των γυναικών, αυτά ίσως θα είναι το αντικείμενο ενός άλλου γύρου συζητήσεων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα μόνο για τα άτομα που έρχονται από Ισλαμικά κράτη σε ό,τι αφορά την παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών. Αυτό είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κύριε Σαντόφσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. με κυρία Επίτροπε, έχω τις εξής ερωτήσεις. Πώς σκοπεύετε να επαναξιολογήσετε το σχέδιο για την ενσωμάτωση των ε, Ευρωπαίων εισαγγελέων στη δομή του Eurojust με μηδενικό κόστος. Και επίσης οι υποθέσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Eurojust είναι όλο και πιο άριθμες. Και θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Άλλη μια ερώτηση, γιατί η ομάδα μου έθεσε το ερώτημα στον κύριο Αβραμόπουλο το σχετικό με τους ε, μαχητές από διάφορες χώρες. Θα ήθελα να υποβάλω από διαφορετική σκοπιά το ίδιο ερώτημα και σε εσά. Δηλαδή, αν Ευρωπαίοι οι οποίοι πηγαίνουν για να πολεμήσουν σε άλλε χώρε όπου υπάρχουν εμπόλεμε καταστάσει και επιστρέψουν κάποια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύετε ότι θα πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη σκοπεύετε να προχωρήσετε στην ανάπτυξη κοινών κατευθυντηρίων γραμμών για τα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτών των ε, ε, ε, πολιτών. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς για την Eurojust. και την ΕΠΠΟ. Θα ήθελα να δηλώσω ότι βεβαίως θα πρέπει να έχει τα μέσα για να αναπτύσσει τις έρευνες και τις ανακρίσεις της Eurojust. Αλλά, ε, όπως ε, πιστεύω, θα πρέπει ε, να στελεχωθεί χωρίς δημοσιονομικές ε, επιπτώσεις. Αυτό που αναφέρεται είναι και η περίπτωση της Όλαφ. το Γραφείο του Ευρωπαίου Δημόσιου Κατήγορου, PPO, θα πρέπει να συνεργάζεται, να έχει την συνεργασία και υποστήριξη της Όλαφ για την καταπολέμηση του εγκλήματος όσον αφορά την οικονομική και εδώ κυρίως ε, θα αναφερθώ στα διαφορετικά ταμεία. Για τη Eurojust λοιπόν πιστεύω ότι είναι δυνατό να στελεχωθεί ε, με μηδενικό κόστος. Θα αναθέσω την εξέταση τέτοιων ε, δυνατοτήτων και αν προχωρήσουμε και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε γιατί οφείλουμε να προχωρήσουμε. Εάν προχωρήσουμε λοιπόν στην θέσπιση μιας δομής για το γραφείο του Ευρωπαίου Δημοσίου Κατηγόρου κατά τρόπον ώστε να έχει και τις τη λειτουργία του σε μελών θα πρέπει αυτό να γίνει και με αντιμετώπιση του κόστους. Θα πρέπει δηλαδή να διερωτηθούμε εάν υπάρξει επιπλέον κόστος, κατά πόσον αυτό ε, υπερκαλύπτει, υπερκαλύπτεται από την προστιθέμενη αξία της ύπαρξης μιας τις υπηρεσίας. Τώρα για τους μαχητές Εδώ έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, μετά επιστρέφουν στη χώρα τους, μα προφανώς αυτοί θα πρέπει να διωχθούν από τη δικαιοσύνη, ωστόσο είναι ζήτημα των κρατών μελών. Αλλά πολύ ε, ευχαριστώ, θα συζητήσω το θέμα αυτό με τον συνάδελφο, τους συναδέλφους που θα έχουν την αρμοδιότητα. Σας πιέζω για το χρόνο, κυρία υποψηφία, γιατί θα πιεστούν αντίστοιχα και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που έχουν ζητήσει το λόγο. Εκ μέρους των Δημοκρατών, η κυρία Σωράια Πόστη παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Γιουρόβα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στοχεύσει στην κοινωνική ενσωμάτωση των Ρωμά. Βλέπουμε όμως τα ακροδεξιά κόμματα να χρησιμοποιούν τα θέματα αυτά ε, στην πολιτική τους εναντίον των Ρωμά. Εμείς έχουμε πάρει αποφάσεις όπως είπα και στα πλαίσια των συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, για την ενσωμάτωση αυτής της κατηγορίας του πληθυσμού. Μήπως θα πρέπει ε, επίσης να ορίσουμε τις, την ρητορική τη βία εις βάρος των Ρωμά σαν κάτι το απαράδεκτο σαν έννοια, κάτι το οποίο θα ενισχύσει τα δικαιώματα των Ρωμά. Και να προσέξουμε σε αυτή την περίπτωση βέβαια και το θέμα της διάστασης ε, των φίλων. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, έρχομαι στο θέμα των Ρώμα, ίσως δεν το έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα αρκετά αναλυτικά. Το θέμα της συμπερίληψης αυτής της, κοινής, της, της κοινωνικής κατηγορίας έχει φυσικά και οικονομικές διαστάσεις. Θα πρέπει φυσικά να ενταχθούν σαν παράδειγμα στην αγορά εργασίας. Δεν μπορώ να μακρηγορήσω, είναι πάντως ένα πολύ περίπλοκο θέμα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα αυτά εναντίον των Ρωμά με διαφορετικό τρόπο μάλλον σε κάθε χώρα μέλος. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπάρξει μία λύση η οποία να είναι καλή για όλες τις χώρες. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική έχει ένα σωστό στόχο και τα κράτη-μέλη πρέπει να παρουσιάσουν τις εθνικές στρατηγικές οι οποίες αντικατοπτρίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διάφορες χώρες. τότε θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και ε, να δούμε ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι ε, σε τομείς όπως η εκπαίδευση, δεν θα τα επαναλάβω αυτά ε, ξέρετε μιλήσαμε για τα ειδικά σχολεία. Ένα άλλο θέμα είναι η κατοικία, ε, είναι η φροντίδα στο σπίτι, όπως επίσης και η αγορά εργασίας. Αυτοί οι τέσσερις τομείς είναι τομείς στους οποίους πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την ενσωμάτωση των Ρωμά. αλλά αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να εξετάσουν κυρίως τα κρατημέλη και φυσικά να το συζητήσουμε και μαζί μας ε, και με, άλλες, ε, και με άλλες, και άλλα επίπεδα εξουσίας όπως οι τοπικές και δημοτικές αρχές. Κύριος Κέρκοπ. Εγώ απογοητεύτηκα από την ερώτησή σας για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Είναι σαφές ότι εμείς επιθυμούμε μεταρρυθμίσεις στον τομέα αυτό. Πώς βλέπετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εσείς το θέμα του σεβασμού των νομικών παραδόσεων, όχι μόνο λόγω των διαφορών ανάμεσα στο αστικό και στο ποινικό κομμάτι, αλλά και για τις χώρες οι οποίες έχουν μεικτά συστήματα. Στον τομέα των διακρίσεων υπάρχει άλλος τρόπος καταπολέμησης των διακρίσεων σε επίπεδο ευρωπαϊκό ε, χωρίς νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. Γιατί οι διακρίσεις ε, εις βάρος των αναπήρων έχει εξαιρεθεί από το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχει τεθεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων ε, που αφορούν τις κοινωνικές υποθέσεις και την απασχόληση. Ευχαριστώ. Λέει υποψήφια επίτροπος. Δεν ξέρω τώρα αν σας κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Καταρχάς μου λέτε ποιες είναι οι διαφορετικές νομικές παραδόσεις. Φυσικά υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο κοινό δίκαιο από τη μία και στο υπηρετικό δίκαιο από την άλλη. Πρόκειται για δύο διαφορετικές παραδόσεις που θα πρέπει να γίνουν σεβαστές. Δεν είμαι βέβαια βέβαια ότι αυτό ερωτήσατε. Τώρα, δεύτερον, έρχομαι στο θέμα της, των διακρίσεων εις βάρος ε, αυτών που έχουν αναπηρίες. Νομίζω ότι έχουμε πάρει κάποια σωστά μέτρα για τη βοήθεια των ανθρώπων αυτών. Και αυτά τα μέτρα καλύπτουν επίσης και το θέμα της πρόσβασης σε υπηρεσίες, όπως επίσης και το θέμα ε, της ε, ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Νομίζω ότι δεν έχουμε ξεχάσει και εξαιρέσει ε, τους ανθρώπους αυτούς και για στα πλαίσια της καταπολέμησης των διακρίσεων έχετε δίκιο βέβαια σε αυτά τα οποία είπατε. Ε, δεν ξέρω αν απαιτούνται πάντα να υπάρχουν ε, νέες νομοθετικές ρυθμίσεις Ίσως μάλιστα κάποιες από τις νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις να μην είναι κατάλληλες γιατί προσπαθούν να εισβάλλουν σε παραδοσιακά νομικά εθνικά πεδία χωρίς αποτέλεσμα. Έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά στο μέλλον γύρω από αυτό. Οι προσπάθειες ε, νομοθετικών ρυθμίσεων μέσω οδηγιών, μέσω κανονισμών είναι ε, κάτι το θεμητό και πρέπει να το κάνουμε και να λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να βελτιώσουμε και τη συνειδητοποίηση των προβλημάτων από την κοινωνία και εδώ ίσως καλούνται να παίξουν σημαντικό ρόλο και οι μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις. Ο κύριος Τσάκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Ρόβα. είπατε ότι οι διακρίσεις δεν πρέπει να έχουν θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, οι αυτόχθονες εθνοτικές μειονότητες, ιστορικές μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αποτελούν 10% όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποια βήματα θα αναλάβετε για να επεκτείνετε την νομοθεσία κατά των διακρίσεων στις αυτόχθονες μειονότητες, ώστε να υπάρξει αποτελεσματική τους προστασία. Δεύτερον, τι μέτρα θα λάβετε για να εξασφαλίσετε ότι έχουν ίσα δικαιώματα και ίση μεταχείριση σε σχέση με τον πλειοψηφούντα πληθυσμό στις χώρες τους και τρίτον ποιες δράσεις θα αναλάβετε έναντι των κρατών μελών που δεν σέβονται τα δικαιώματα των εθνοτικών μειονοτήτων και κάνουν διακρίσεις εναντίον τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσάκα για το ερώτημά σας. Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το θέμα αυτό με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Βιέννη. που είναι ο φορέας πιστεύει ότι αυτό είναι πράγματι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιληθεί και με ρωτάτε τι θα κάνετε πρώτα απ' όλα. Θα προσπαθήσω να αναλύσω τα δεδομένα και τις στατιστικές που έχουμε και τις μελέτες που έχουμε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι μειονότητες σε διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχουν διαφορετικές προσέγγισεις στα κράτη-μέλη έναντι των μειονοτήτων. Αυτή τη στιγμή δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία αλλά πιστεύω ότι οι εθνοτικές μειονότητες καλύπτονται από όλε τις πρόνοιες που προστατεύουν άτομα και πολίτες εναντίον οποιασδήποτε μορφής διάκρισης. Επομένως η προστασία που έχουν είναι η ίδια προστασία που έχουν άλλες μειονοτικές ομάδες του πληθυσμού σε σχέση τώρα με την εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τα εργαλεία και τα μέσα ώστε να αναλάβει δράση εάν ένα κράτος μέλος δεν σέβεται τα νομικά, τις νομικές πρόνοιες και διατάξεις των συνδικών. Έχουμε λοιπόν όλες αυτές τις διαδικασίες που θα μας επιτρέψουν να αναλάβουμε δράση. Αλλά δεν μπορώ τώρα να είμαι πιο συγκεκριμένη. Και δεν θεωρώ ότι έχω στοιχεία για τέτοιες παραβιάσεις. Για την ε, ομάδα των Σοσιαλιστών, ο κύριο Λοπέ Φερνάντο Αγγιλάρ, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Λίμπερ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, εδώ είμαι. Κυρία υποψήφια επίτροπε, καλώ ήλθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην ακρόαση αυτή και στο γύρο ερωτήσεων της Λίμπε. Νομίζω ότι είχατε εκφράσει καταρχήν ενδιαφέρον για το χαρτοφυλάκιο της εσωτερικής αγοράς, αλλά η δικαιοσύνη και η ισότητα των φύλων δεν είναι ίσον χαρτοφυλάκιο. Ίσα ίσα είναι μια από τις πιο σημαντικές ε, εκφάνσεις, πολιτικές εκφάνσεις του συνταγματικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ε, ασφάλεια, δικαιοσύνη και ελευθερία και με την ε, συνεργασία των νομικών υπηρεσιών και των συστημάτων δικαίου και του εισαγγελέω για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά είναι θέματα που είναι πάρα πολύ κέρια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να υπάρξει λοιπόν νομοθεσία για τα θέματα αυτά και η ενθρόνηση ενό δημοσίου εισαγγελέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ποιε είναι λοιπόν οι απόψει σα για την θέση του Συμβουλίου για τον κανονισμό που θα θεσπίσει το γραφείο της εισαγγελίας, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεύτερον, πώς θα εξασφαλίσετε την πρόοδο για την διαδικασία του πακέτου που έχει να κάνει με τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων. Και τρίτον, πώς θα εξασφαλίσετε ότι οι αρμόδιοι φορείς μεταξύ των οποίων το Eurojust, το Europol και το γραφείο του Ισαγγελέως καθώς και η Όλαφ θα συνεργάζονται και θα δρουν με τρόπο ο οποίος συνάδει με την Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. έχει τρεις ε, τεράστιες πτυχές στο ερώτημά σας και λόγω του χρόνου θα περνάμε σύντομη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προβλέπεται από το άρθρο 86 των συνθήκων που ζητά την δημιουργία αυτού του θεσμού ώστε να εξασφαλιστούν τα συμφέροντα των Ευρωπαίων φορολογουμένων και να αντιμετωπιστεί το θέμα της διαφθοράς και της απάτης κατά του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Είναι λοιπόν ένα δύσκολο. Ε, είναι πολύ δύσκολο να αγνοήσει κανείς αυτό το θέμα το οποίο είναι σαφώς καθαγιασμένο στην ε, συνθήκη. Βέβαια δεν αμφισβητεί κανείς τον θεσμό αυτό του, της εισαγγελία, αλλά είναι διαφορετικό το να μπορέσουμε να βρούμε τη συγκεκριμένη διασύνδεση του γραφείου αυτού της εισαγγελία και των εθνικών εισαγγελικών αρχών. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο θα χρειαστούμε μια μακρά διαδικασία διαλόγου σε τεχνικό επίπεδο για τη σωστή κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ του Ευρωπαίου Εισαγγελέα και των Εθνικών Εισαγγελέων και φυσικά δεν νομίζω ότι έχω το χρόνο τώρα να μπω σε το θέμα αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν το δεύτερο ερώτημα γιατί δεν μπορώ να διαβάσω τις σημειώσεις μου. Αλλά παρόλα αυτά η συνεκτικότητα των δράσεων των διαφορών φορέων και της εφαρμογής του ποινικού δικαίου. Όλα αυτά που θα κάνουμε λοιπόν για την εισαγγελική αρχή ήδη απαιτούν καλή συνεργασία του Europol, Eurojust, του Olaf, της Olaf και του εισαγγελέα. Νομίζω λοιπόν ότι ο νέος κανονισμός που είναι σε κατάσταση προσχεδίου για την ΟΛΑΦ ε, σίγουρα παρατρύνει όλους αυτούς τους θεσμούς σε συνεργασία. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν το δεύτερο ερώτημά σας. Εντάξει, είναι τα ε, δικονομικά δικαιώματα των κατηγορουμένων και των υπόπτων. Εγώ συμφωνώ με τι προτάσει που έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα, τόσο σε ό,τι αφορά το τεκμήριο αθωότητο, όσο και την παροχή νομική βοήθεια και τα δικαιώματα των παιδιών. Δεν έχω κανένα επιχείρημα εναντίον όλων αυτών. Σα ευχαριστούμε για την απάντηση και στο τελευταίο ερώτημα, λέει ο κύριο Μωράης. Θέλω να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος όλων των μελών τη Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων και θα δώσω τώρα το λόγο μετά από κάποια ε, χορογραφία μεταξύ των ε, Προέδρων των Επιτροπών στον πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικής, στην πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς. Well, there's no time, Oh, no, no, it can go over two hours. It's, no, it's a minimum. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα προεδρεύουν οι γυναίκες, κυρία Γεωρούβα. για να συστήσουμε θέματα εσωτερικής αγοράς και θεμάτων των καταναλωτών. Όπω ξέρετε αυτή η Επιτροπή Ιστορική αγορά και Θεμάτων Καταναλωτών έχει σαν ρόλο την προστασία τη ορθή λειτουργία τη ιστορική αγορά και την αποδιάρθρωση φραγμών στη λειτουργία αυτή, συμπεριλαμβανομένη και τη ψηφιακή αγορά, και ιδιαίτερα όσον αφορά το ρόλο ε, με ρημνά ιδιαίτερα για την προστασία και προαγωγή των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, καθώ και θέματα νομοθεσίες που έχουν να κάνουν με την επιβολή και τήρηση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς και των ε, δικαιωμάτων των καταναλωτών στόχων της συνάντησης αυτής είναι να αντιληφθούμε τις δικές σας θέσεις στους συγκεκριμένους αυτούς τομείς για να ε, αντιληφθούμε πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις τομείς αυτούς. Η Επιτροπή μας στόχο έχει να κοιτάξουμε πιο συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε λειτουργικό επίπεδο που ε, μεταφέρθηκαν από το το αρμοδιοτήτων σε άλλου, ε, σε θέματα που αφορούν το των καταναλωτών. Και τώρα περνάω στην, κυρία, στην πρώτη ερώτηση με την κυρία Μετσόλα, εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ξεκινώντα να συμφωνήσω με τον Τίμωθη Κέρκοπ όταν είπε ότι δεν θα έχετε ιδιαίτερη, θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα των ανθρώπων με αναπηρία Θα ήθελα ωστόσο να ε, επικεντρωθώ στις, ε, στους ιστοτόπους Προφανώς θα πρέπει στο θέμα αυτό να αποτραπούν οι καταχρήσει, θα πρέπει ο πολίτης να τοποθετηθεί στο επίκεντρο της χάραξη πολιτικής. Ερωτήσεις λοιπόν, εφόσον επί στι θέσει του Πιτρόπου σκοπεύετε να μεριμνήσετε ώστε να δημιουργηθούν τα μέσα αυτά και τι μέτρα σκοπεύετε να αναλάβετε για τον εξορθολογισμό και την ορθή λειτουργία αυτών των ιστοτόπων, κάποιο σύστημα πιστοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα βοηθήσει τον καταναλωτή να εντοπίσει ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι παίζουν σωστά του όρου του παιχνιδιού. Ε, για την ε, διαγραμμική επίλυση διαφορών βλέπετε δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερων πόρων ώστε να εξασφαλίσετε και η μετάφραση. Ευχαριστώ. Παρακαλώ για την απάντηση. Σας ευχαριστώ. Το διαδίκτυο σε ευρία έννοια είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να οδηγήσει και σε παραπληροφόρηση ακόμη και να παρασύρει ε, ευάλωτες ομάδες πληθυσμού σε λάθος επιλογές. Μπορεί να πέσουν θύματα απάτης ε, μπορεί να παρασυρθούν από ε, παραπληροφόρηση, από σφαλμένη ενημέρωση, θεωρώντας ότι κάτι μπορεί να προσφέρεται δωρεάν, ενώ ε, πέφτουν στην παγίδα και αγοράζουν προϊόντα το ένα μετά το άλλο και εδώ αναφέρομαι παραδείγματι στα παιδιά που χρειάζονται προστασία από τέτοιου είδους απάτες αλλά και ηλικιωμένους που δεν είναι σε θέση πάντοτε να αξιολογούν τις πληροφορίες με την ίδια ευχέρεια. Πρέπει λοιπόν να μεριμνούμε ώστε να μην επιτρέπεται στους ιστοτόπους να διαδίδουν, να, παρουσιάζουν εσφερμένες πληροφορίες, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να μεριμνούμε ώστε αυτήν ό,τι δηλώνουν είναι σαφές και ξεκάθαρο. Υπάρχουν λοιπόν αρμόδια εθνικά όργανα ε, εποπτείας του διαδικτύου, τα οποία θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να ε, αποτρέπονται αυτές οι αθέμητες πρακτικές. Το πώς θα γίνει αυτό συγκεκριμένα δεν μπορώ να σας το ε, πω, διότι δεν έχω μελετήσει το θέμα αυτό. Για τις μεταφράσεις και τα σχετικά κονδύλια πρόκειται για ένα ουσιώδες ζήτημα και θα χρειαστεί να το συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα να ε, δούμε το θέμα της διαγραμμικής επίλυσης διαφορών. Όπως άλλωστε και με το θέμα της, ε, του χώρου ηλεκτρονικής δικαιοσύνης θα πρέπει να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση ώστε να εξασφαλίζει ο ενδιαφερόμενος τη μετάφραση στη μητρική του γλώσσα. Βεβαίως ε, ε, θα αναλάβω τη σχετική δράση εφόσον λάβω και τα καθήκοντα αυτά, αλλά βλέπω ότι έχω ξετλήσει τον χρόνο μου. Κυρία Γκέπχαρτ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Υποψήφια Επίτροπε έχετε αρμοδιότητα σε ένα τεράστιο θέμα προστασία του καταναλωτή που έχει μια ε, διάσταση και εγκάρσια και αγγίζει ως εκ τούτου πολλούς άλλους τομείς. Ε, αυτές τις αρμοδιότητες με την εγκάρσια προσέγγιση πώς σκοπεύετε να τις αναπτύξετε στους επιμέρους τομείς αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτη ερώτηση επιπλέον. Θα ήθελα να επισημανώ ότι έχω ακούσει κάπως αντιφατικό θετικές ειδήσει και φήμες, μάλλον απαντήσεις από πλευρά σας για το πώς σκοπεύετε να χειριστεί το θέμα των καταναλωτών. Φέρει ε, ε από τις τιμής στο καταναλωτικό δίκαιο λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα, ε, ένα δίκαιο για τους καταναλωτές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε κράτους ενώ από την άλλη είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο δίκαιο για τους καταναλωτές, ένα πραγματικά ενιαίο. Ε, τι θέλετε εν τέλει. Τι είδους νομοθεσία για τα δικαιώματα του καταναλωτή και την προστασία του καταναλωτή θέλετε στην Ευρώπη. Απάντηση. Ευχαριστώ. Η κατανάλωση των καταναλωτών δεν είναι η μόνη εγκάρση αρμοδιότητα που έχω στο χαρτοφυλάκιό μου. Αλλά τώρα θα ήθελα να αναφερθώ ε, πολύ πιο συγκεκριμένα για να ε, διασκεδάσω κάποιες ανησυχίες ότι υπάρχει κίνδυνος να παραμεληθεί το θέμα αυτό από το χαρτοφυλάκιό μου. Κοιτάξτε, καταναλωτές είμαστε όλοι. Όλοι εμείς που καθόμαστε εδώ είμαστε καταναλωτές. Ο καταναλωτής έχει τεράστια ε, ισχύ και αν οι στατιστικές που έχω στα χέρια μου αληθεύουν, έχουμε το 56% του ΑΕΠ στα χέρια του καταναλωτή. Άρα η ενίσχυση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή έχει κρίσιμη σημασία. Η δραστηριοποίηση του καταναλωτή έχει ρόλο κινητήριου μοχλού για την οικονομία και την κοινωνία και αυτά δεν είναι λόγια απλώς έχουν τεράστια σημασία στην πράξη και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να το δει και η Επιτροπή. Αυτό είναι κάτι το οποίο στο συλλογικό όργανο που ονομάζεται Επιτροπή θα φροντίσω να ε, συζητηθεί πολύ συγκεκριμένα και στις οικονομικές χρηματοπιστωτικές ε, δραστηριότητες και οπουδήποτε αλλού πρέπει να υπάρξει εκπροσώπηση του καταναλωτή ε, και να ακουστεί η φωνή του και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε τη θέση των καταναλωτών. Για δε σύγκρουση σχετικά με το ενιαίο δίκαιο των πωλήσεων και την προστασία των καταναλωτών. Σύγκρουση πραγματικά δεν υπάρχει. Το ενιαίο δίκαιο των πωλήσεων ελπίζουμε ότι θα είναι η πρώτη επιλογή για τον πολιτή. Δεν μπορούμε απλώς να περιμένουμε να επιλέγεται μόνο γιατί είναι πιο καλό για τον καταναλωτή, πιο συμφέρον για τον καταναλωτή. Ελπίζουμε ότι το νέο δίκαιο των πωλήσεων θα προτιμηθεί και γιατί προστατεύει τον καταναλωτή, αλλά και γιατί ε, μειώνει το κόστος για τον πολιτή ή μη τι άλλο. Άρα είμαι αισιόδοξη σε αυτό. E Ο κύριος Τίζα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αναφερθήκατε στη, στο νέο πακέτο μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Έχω ένα ερώτημα <clears throat> συγκεκριμένα. Με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσετε ότι αυτές οι αρχές θα εφαρμοστούν στην, ε, στο πακέτο αυτό και επίσης για τα δικαιώματα των καταναλωτών ιδίως όταν αγοράζουν στο ίντερνετ. Τι θα κάνετε για την αναζήτηση, για την ε, αναζήτηση διευθύνσεων IP ε, του διαδικτύου από τις εμπορικές ιστοσελίδες προς εμπορική χρήση και τι θα κάνετε με την πρόσβαση δεδομένων για τομείς πρόσφατα δεδομένα για τομεί που είναι κέρδη, όπω είναι ο τομέα της ε, υγείας και πώ θα εξασφαλίσετε την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα αυτό. Εξάλλου έχουμε την Ευρωπαία Πρωτοβουλία για του πολίτε, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη δημοκρατία τη Ευρώπη. Αυτό το εργαλείο δημιουργήθηκε με αυτόν τον σκοπό. Εδώ θα ήθελα να θέσω το ερώτημα πώ μπορείτε να επηρεάσει αυτό το εργαλείο την ε, δικαιοσύνη, δεδομένου ότι αυτή η πρωτοβουλία πολιτών έχει απορριφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. να ξεκινήσω με την πρωτοβουλία πολιτών. Είναι πράγματι μια μεγάλη επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η δυνατότητα υποβολής πρωτοβουλειών πολιτών και αυτό είναι μια ε, έκφραση της άμεσης δημοκρατίας. Το υποστηρίζω λοιπόν αυτό. Πώς τώρα θα προστατέψουμε τους καταναλωτές από την, ε, από την καταγραφή των ε, δεδομένων τους στο, διαδίκτυο. Η μεταρρύθμιση για τα δεδομένα, των, ε, τα προσωπικά δεδομένα, έχει ένα σημαντικό στόχο. Συγκεκριμένα το να μπορέσει να αυξήσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων ώστε να εμπιστεύονται τους ε, συναλλασσόμενους με αυτούς τις ε, επιγραμμικές συναλλαγές και επομένως να είναι έτοιμοι να δώσουν τα στοιχεία τους, ξέροντας ότι αυτά τα στοιχεία δεν θα τύχουν κατάχρησης για λόγους ε, ασφαλ... ασφάλειας ή για λόγους εμπορικούς. Αυτό είναι λοιπόν προαπαιτούμενο για να εξασφαλιστεί αυτή η εμπιστοσύνη και αν θέλουμε να αυξήσουμε φυσικά τον αριθμό των επιγραμμικών συναλλαγών στο διαδίκτυο. Αυτό λοιπόν είναι και ένας από τους κύριους στόχους της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να προστατέψουμε λοιπόν τους καταναλωτές και αυτό είναι ένα από τα οριζόντια θέματα το οποίο θα αντιμετωπίσει ο κύριο Σέτιγκερ, ο κύριο Σάνσιπ και άλλα μέλη της Κομισιόν, μέλη της Κομισιόν. Φυσικά εγώ πάντα θα υποστηρίξω οποιαδήποτε τέτοια προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων. Κύριο Τσάντσόβερ, από, Τσάντσόβερ από τους φιλελεύθερους. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Για την κυρία Γιάουροβα λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια τεράστια εκστρατεία για την συνειδητοποίηση της σημασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Βασίζεται σε μια μελέτη η οποία δείχνει ότι οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους σωστά. Ιδιαίτερα γύρω από τα θέματα των αγορών μέσω του διαδικτύου σαν η Επίτροπος που θα είσαστε αρμόδια για τον τομέα αυτό, τι μπορείτε να κάνετε έτσι ώστε να κατανοήσουν τη σημασία των δικαιωμάτων τους οι καταναλωτές. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έτσι ώστε να κατανοήσουν τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν και πώς θα αποκαταστήσετε την ισορροπία ανάμεσα στους καταναλωτές από τη μία και στις επιχειρήσεις από την άλλη.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 για την Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω για μια ακόμη φορά στην ερώτηση της κυρίας Γκέπχαρτ που δώσατε στην ε, κυρία Γκέπχαρτ η απάντηση δεν ήταν πλήρης. Λέτε ότι από τη μία θα βοηθήσετε τους καταναλωτές από την άλλη λέτε και στις γραπτές απαντήσεις ότι θέλετε να υπάρξει ισότιμη αντιμετώπιση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Αν εγώ ε, αγοράζω από το διαδίκτυο, ε, έχω τη δυνατότητα να γνωρίσω την νομοθεσία, την καθημερινή η οποία ε, καλύπτει τη συναλλαγή. Αυτό πρέπει να ισχύει με τον ίδιο τρόπο για το σύνολο της Ευρώπης. Βέβαια από την άλλη θα ε, δίνεται τη δυνατότητα στην επιχείρηση να αποφασίζει ε, για το, ε, για το σύστημα το νομικό το οποίο θα καλύπτει νομικά την συναλλαγή. Πρέπει νομίζω να καταλάβετε με αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορείτε ταυτόχρονα να προστατεύετε και τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Eh, děkuji. Eh, já eh, mě mrzí, že působila moje odpověď zmatečně. Já se to zkusím. ίσως ε, πράγματι να δημιούργησε μία κάποια σύγχυση η απάντηση την οποία σας έδωσα θα την επαναλάβω. Όπως είπα εγώ θα προασπιστώ τα συμφέροντα των καταναλωτών. Θα προσπαθήσω έτσι ώστε οι καταναλωτές που είναι ο ασθενής συναλλασσόμενος, αν θέλετε, στα πλαίσια μιας συναλλαγής να προστατεύεται σωστά. Να είναι σωστά ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους και στα πλαίσια του νέου ευρωπαϊκού λεγόμενου νόμου για τις πωλήσει. Θα υπάρχει η δυνατότητα λοιπόν χρήσης του νομικού καθεστώτος αυτού του νέου νόμου ε, εναλλακτική σε σχέση με τις εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις. αν μια επιχείρηση ε, ε, ασκεί τις εμπορικές της δραστηριότητες διασυνοριακά είναι κάτι το οποίο λειτουργεί θετικά για αυτήν την επιχείρηση και θα έχει την δυνατότητα επιλογής του συγκεκριμένου νομικού καθεστώτος να μην ξεχνάμε ότι οι νομικές ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι φυσικά υποφελείς όχι μόνο για τον επιχειρηματή αλλά και τον καταναλωτή. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχουν προβλέψεις οι οποίες μπορεί να λειτουργήσουν σωστά και για τις δύο πλευρές. Ο επιχειρηματικός κόσμος κατανοεί ότι ο ικανοποιημένος καταναλωτής είναι αυτός ο οποίος θα επανέλθει και θα αγοράσει περισσότερες, ε, περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες. Συνεπώς δεν υπάρχει αντίφαση σε αυτά τα οποία λέμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκ, των, μέρους των Πρασίνων ο κύριος Άρμπρεχτ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γιώργοβα, σας ευχαριστώ για τις τοποθετήσεις σας μέχρι τώρα, ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για μένα είναι πολύ σημαντικό ο στόχος αυτός, τον οποίο έχετε καταγράψει στις γραπτές σας ε, ε, απαντήσεις για μια έγκριση του πακέτου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσα στο προσεχής εξάμεινο να είναι και ρεαλιστικός. Το πρόβλημα είναι ότι τώρα, ε, εάν δεν κάτσουμε στο τραπέζι να διαπραγματεύσουμε με το Συμβούλιο των Υπουργών, δεν θα φτάσουν αυτοί οι έξι μήνες. Επιτάπητος βρίσκονται δύο θέσεις, μία του Κοινοβουλίου, μία του Συμβουλίου και πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση. Ε, ο τριμερής διάλογος να ολοκληρωθεί μέσα σε έξι μήνες μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Ρωτώ λοιπόν τι σκοπεύετε να κάνετε έτσι ώστε τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του έτους το Συμβούλιο να καταλήξει να ε, διατυπώσει τις δικές του θέσεις και πάνω απ' όλα να καταλήξει θέσει θέσεις οι οποίες δεν θα απέχουν τόσο πολύ από αυτές τις δικής μας θέση του Μαρτίου. Απάντηση. Ευχαριστώ. Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τα όσα έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εσείς προσωπικά, κύριε Άρμπρεχτ. Γιατί μας βοήθησαν να προχωρήσουμε Όντως, ε, περνάει πολύ γρήγορο ο χρόνος, το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι πολύ πιεστικό. Πρέπει όμως να τηρηθεί και να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα παρά τη δυσκολία στις ε, διαπραγματεύσεις. Ξέρω ότι υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο το σύστημα προστασίας των προσωπικών δεδομένων μπορεί να αποδειχθεί λειτουργικό, φοβούνται μήπως ε, επιβάλλει υπερβολικό γραφειοκρατικό βάρος ε, για τις αρχές διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Ξέρω ότι είχατε διατυπώσει κάποιες ε, προτάσεις και εσείς όσον αφορά το νόγκο των δεδομένων που θα μπορούσαν να υπαχθούν στο σύστημα αυτό. Επομένως, αφενός μεν προσπαθούμε να περιορίσουμε την επιβάρυνση, τη γραφειοκρατική, ε, την πρακτική, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ε, εξασφαλίσουμε και τις ελάχιστες προϋποθέσεις. Πρέπει να δούμε τι μπορούν να κάνουν και οι εταιρείε βέβαια και η ευελιξία. Η ευελιξία ως προς την διαχείριση ε, από τους δημόσιους φορείς των προσωπικών δεδομένων έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν τις προϋποθέσεις και τις διτυπώσεις για τις δημόσιες αρχές. Εδώ ε, υπησέρχονται πολλά και τεχνικά ζητήματα, αλλά και αισθήματα ουσίας. Θα πρέπει λοιπόν ε, να μην ότι ο τελικός στόχος είναι το υποχρεωτικό αποτέλεσμα, δηλαδή η ε, αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε μια οδηγία του 1995. Ευχαριστώ εκ μέρους της Ευρώπη των Ελευθεριών και των Δημοκρατιών, Ταϊάν Τζέιμ. Ευχαριστώ. Υποψήφια, κυρία Επίτροπε, στο Ηνωμένο Βασίλειο περιμένανε ότι ο Λόρδο Χίλ θα αναλάβει το θέμα των ε, πόνου των τραπεζικών στελεχών. Αλλά τώρα μάθαμε ότι έχει περάσει στο δικό σα χαρτοφυλάκιο μεταξύ των άλλων θεμάτων των καταλωτών. Τρία ερωτήματα εδώ. <clears throat> Θεωρείτε και συμφωνείτε ότι το να περιορίζει κανεί τα μπόνους σε μια ανταγωνιστική αγορά θα οδηγήσει σε υψηλότερου μισθούς. Δεύτερον, συμφωνείτε ότι με το να αυξήσετε το πάγιο κόστο μιας επιχείρησης αυξάνεται την πιθανότητα να πτωχεύσει. Και τρίτον, σε οποιαδήποτε περίπτωση αναδιαπραγμάτευσης θα υποστηρίζατε την αίτηση του Ηνωμένου Βασιλείου να εμποδίσουν τους ε, Ευρωκράτες και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να επεμβαίνει σε ιδιωτικού χαρακτήρα συμβάσεις. Ευχαριστώ για το ερώτημά σας. Πρώτα απ' όλα, θέλω να πω ότι η εποπτεία των πόνους των τραπεζικών σε σχέση με τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν είναι κάτι το οποίο για μένα είναι κάτι το οποίο είναι μια σωστή αρχή. Εγώ πιστεύω ότι οι κανόνες πρέπει να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξει δυνατότητα ηθικού κινδύνου για τα τραπεζικά στελέχη και να μην αναλαμβάνουν κινδύνους μονάχα με βραχυπρόθεσμη οπτική γωνία. Θα πρέπει να παραεμποδίσουμε επίσης οποιαδήποτε παραβίαση και ζημιά στα δικαιώματα των μετόχων, αλλά επίσης και του γενικού κοινού. Ξέρουμε ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να έχει επιρροή στην γενικότερη οικονομία. Για τα ερωτήματα τώρα που θέσατε, αν αυτή η μείωση των πόνους μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των ε, αποδοχών και αν μπορεί να οδηγήσει η αύξηση του κόστου σε πτώχευση επιχειρήσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχω μελετήσει και πιστεύω μετά από αυτά που έχω μελετήσει μόνο 1% των εργαζομένων καλύπτεται από αυτό τον περιορισμό στα μπόνους και είναι αυτοί οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τις ε, επενδύσεις κινδύνου. <clears throat> αυτό λοιπόν δεν είναι τόσο κέριο θέμα όσο αφορά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Εγώ δεν μπορώ να κρίνω το ευρωπαϊκό, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η πρώτη ε, η διαδικασία έλαβε χώρα στις 8 Σεπτεμβρίου και περιμένουμε την οριστική απόφαση του δικαστηρίου μέχρι το τέλος του χρόνου. Και στη συνέχεια εμείς θα πρέπει να εφαρμόσουμε την απόφαση και θα δούμε τι μεταρρυθμίσεις πρέπει να προκύψουν. Φυσικά θα προκαταλάβω τη δικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο κύριος Πόσπισιλ. Καλησπέρα σας κυρία Γιώργο. Θα ήθελα να πω πρώτα ότι τα σχέδια της Επιτροπής για την ε, αξιολόγηση της ευρωστίας και της λειτουργικότητας της ισχύουσας νομοθεσίας θα οδηγήσουν την Επιτροπή σε πιθανή συγχώνευση, κωδικοποίηση κανόνων ε, για το προσωπικό των καταναλωτών, τη διαφήμιση κτλ. Εγώ λοιπόν θα αναφερθώ στο δίκαιο των καταναλωτών και θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα οράματά σας τα σχετικά με πιθανές αλλαγές σε ποιους τομείς θα θέλατε να επικεντρωθείτε. Και σε σχέση με τις αθέμητες πρακτικές στις βάρος των καταναλωτών ή με τις αθέμητες συνθήκες που ε, περιέχονται σε συμβάσεις, ε, τι μπορείτε να κάνετε. Ευχαριστώ. Όπως ε, ανέφερα και νωρίτερα, έχουμε να κάνουμε την οδηγία για την προστασία των καταναλωτών. Πολύ καλό είναι να προτείνονται νέες νομοθετικές προτάσεις, μερικές φορές όμως μπορεί και λόγω των κατευθυντηρίων λόγω και των χρονοδιαγραμμάτων που είναι πιεστικά, είναι σκοπιμότερο να επικεντρωνόμαστε στην ορθή εφαρμογή των εφαρμοζομένων κανόνων. Για δε τις αθέμητες πρακτικές, ε, υπενήσεστε πρακτικές της ε, τσεχικής δημοκρατίας, στην τσεχική δημοκρατία, όντως είχαμε μια πολύ δυσάρεστη υπόθεση κατάχρησης εμπιστοσύνης ηλικιωμένων πολιτών, με στόχο την εξαπάτηση, τους προσκαλούσαν σε διάφορες εκδηλώσεις όπου αναγκάζονταν να αγοράζουν διάφορα προϊόντα. Αυτό είχε και τραυματικές ακόμη συνέπειες, για να μην μιλήσω για τις οικονομικές συνέπειες. Βεβαίως λοιπόν και είμαι κατά των ε, πρακτικών αυτών, βεβαίως και είμαι υπέρ της καταπολέμησης τους, της καταπολέμησης της παραπραγματικής διαφήμισης. Και επίσης θα πρέπει πιστεύω να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί ε, το κείμενο της οδηγίας για την ασφάλεια των προϊόντων και για την ε, παρακολούθηση της λειτουργίας της αγοράς, εποπτεία στην αγορά. Αυτά είναι τα δύο κύρια νομοθετήματα και πιστεύω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε τον πολίτη, να θέσουμε τον πολίτη στο επίκεντρο όταν χαράσουμε πολιτικές για τον καταναλωτή. Τον πολίτη που είναι ευάλωτος, και άρα θα ήθελα να γίνει πρώτα μια ανάλυση, μια μελέτη η οποία θα μας δείξει πώς διάφορες ομάδες ευάλωτων πολιτών μπορεί να επηρεάζονται. Και στη συνέχεια μπορούμε να εκδώσουμε τις νομοθετικές προτάσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Σεχνάλοβα. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητή κυρία Γιώουροβα, εδώ είμαι, με βλέπετε. Στα αριστερά σας. Καλώς ήρθατε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη θέση του και πρώτη ανάγνωση για τα θέματα της ασφάλειας των προϊόντων και την επιοπτία της αγοράς. Εφέτος τον Απρίλιο. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για το θέμα αυτό που έχει τόση σημασία για τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Δυστυχώς όμως το θέμα αυτό παρακολύεται σε επίπεδο Συμβουλίου. Όπως γνωρίζετε το κύριο κόλλημα είναι το άρθρο 7 για την ρήτρα Made In εσείς ε, αναφερθήκατε στο θέμα αυτό και θέλω να σας ρωτήσω πώς μπορείτε να βοηθήσετε για την αντιμετώπιση του αδιεξόδου σε επίπεδο Συμβουλίου. Και πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, πώς μπορείτε λοιπόν να βοηθήσετε στην αντιμετώπιση του και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το ε, πρόβλημα της ρήτρας. Ε, για το Made in του άρθρου 7. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Σεχνάλοβα. Η προαγωγή της οδηγίας αυτή για την προσθέτωση του καταναλωτή είναι μια από τις μου και ας μην το τόνισα τόσο. Ε, νομίζω ότι έχει γίνει αρκετή δουλειά ήδη και θα ήταν κρίμα, θα ήταν πολύ λυπηρό να χρειαστεί να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια αυτή για ένα άρθρο που το οποίο βέβαια συμφωνώ είναι πολύ σημαντικό. Τώρα θα κάνω κάτι τώρα που ίσως να μετανιώσω μετά, αλλά θα σας ε, προτείνω τρεις διαφορετικές επιλογές και ελπίζω να μην διαγνώσετε από τα λόγια μου αυτήν που προτιμώ προσωπικά. Γνωρίζω λοιπόν ότι δεν έχει γίνει μελέτη αξιολόγησης των συνεπειών της, ε, του άρθρου 7. Έχουν γίνει πολλές προτάσεις σε αυτό. Μπορούμε να αναλάβουμε μια τέτοια πρωτοβουλία, δηλαδή μπορεί να γίνει μια αξιολόγηση του σε ποιο βαθμό ε, η ετικέτα ε, made in μπορεί να αλλάζει την, ε, τις συνθήκες σχετικά με ένα προϊόν για να δούμε και τα θέματα της ασφάλειας. Άρα μπορούμε να κάνουμε πρώτα την αξιολόγηση και μετά να αρχίσουμε να συνομιλούμε πάλι με τα κράτη-μέλη για το εάν είναι καλή η πρόταση του ΜΕΙΝΤΙΝ ή όχι και ποια είναι η μορφή με την οποία ε, μπορεί να υιοθετηθεί αυτή η ρήτρα ή αυτή η ετικέτα. Μια άλλη λίστα ήταν το άρθρο 7 να διαγραφεί. Υποθετική περίπτωση πάλι, γιατί πιστεύω ότι θα προκύψει τεράστια αντίδραση, εξάλλου δεν πρόκειται για αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τρίτη επιλογή, η απόσυρση της προτάσεως. Ε, κάτι το οποίο θα ήθελα οπωσδήποτε να αποφύγω, γιατί πρόκειται για ένα νομοθέτημα αναγκαίο, για ένα νομοθέτημα στο οποίο έχει γίνει ήδη πάρα πολύ δουλειά. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει πρώτα μια αξιολόγηση επιπτώσεων και μετά να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει με τα κράτη-μέλη. Τελευταίος. Τελευταία ερώτηση από τον κύριο Ροσφόρ. Ευχαριστώ κυρία Γιαούροβα. Σας ευχαριστώ και για τις δηλώσεις σας υπέρ των καταναλωτών. Ευχαριστώ και για τις προτεραιότητές σας. Είναι σπάνιο μια πολιτική υπεύθυνη να προέρχεται από τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Ελπίζω αυτό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τις στάσεις και τις αντιλήψεις των πολιτών και των καταναλωτών. Ε, να γίνω πιο συγκεκριμένος. Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Διαδικτυακής Επίλυσης Διαφορών. Αναφερθήκατε σε αυτό. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Ήδη στις 9 Ιουνίου του 2015 οι υπηρεσίες σας θα πρέπει να διασφαλίσουν τις γλωσσικές υπηρεσίες τις οποίες αναφερθήκατε στο φιλικό χαρακτήρα της πλατφόρμας κτλ. Έχει σημασία αυτό για μας ε, στην Επιτροπή μας, στην ΙΜΚΟ, γιατί θεωρούμε ότι η προάσπιση των καταναλωτών είναι νομικό θέμα, μεν, αλλά ό,τι έχει σχέση με την διαιτησία και το εξοδικαστικό κομμάτι είναι κάτι που πρέπει να δοκιμαστεί σωστά. Ευχαριστώ. Και εδώ έχω συγκεκριμένες ε, αναμνήσεις προσωπικές γιατί όταν ήμουν υπουργό εν περιπτώσει είχαμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό της δυνατότητας δημιουργίας μιας πλατφόρμας για την επίλυση των διαφορών των εμπορικών. Γι' αυτό λοιπόν θέλω το σύστημα να είναι αποτελεσματικό, να είναι ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται και να μην είναι μια πραγματικά φρούδα επένδυση. Ε, ελπίζω ότι το σύστημα εν πάση περιπτώσει θα λειτουργήσει σωστά και θα προτιμηθεί από τους χρήστες και τους πολίτες, τους απλούς πολίτες και τους επιχειρηματίες. Ελπίζω επίσης ότι το σύστημα το οποίο στην παρούσα φάση βρίσκεται σε ε, δοκιμασία δειγματοληπτικά επελέγησαν ορισμένοι χρήσεις, αλλά θα πρέπει να τεθεί σε πλήρη λειτουργία από τα μέσα του 2015. Αυτή είναι η υποχρέωση λοιπόν την οποία κανονικά δεν θα έπρεπε να αναλάβω εδώ, αλλά να πω ότι ήδη από τις αρχές του 2015 το σύστημα θα είναι λειτουργικό, θα είναι διαθέσιμο για ε, διαδικασίες ε, επίδειξης λειτουργίας και σε τεχνικό επίπεδο μας έχουν διαβεβαιώσει ότι το σύστημα θα είναι επίσης διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης της επίσημης. Ελπίζω λοιπόν όλα να πάνε καλά και από τον επόμενο χρόνο να μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε επίσημα το σύστημα αυτό. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας, για τα ερωτήματα της Επιτροπής ΙΜΚΟ. Τώρα θα περάσουμε στην Επιτροπή ΦΕΜ. Λυπάμαι που καθυστερήσαμε λιγάκι, αλλά θα πάρουμε όλες τις ερωτήσεις από την Επιτροπή ΦΕΜ. Θα προχωρήσουμε λιγάκι περισσότερο μέσα στον χρόνο. Σας ευχαριστώ κυρία Φόρτ, κυρία Γιώουροβα. Δυστυχώς Αυτό το τελευταίο μπλοκ ερωτήσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Η ισότητα των φύλων είναι πάρα πολύ σημαντική στην Ευρώπη. Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να ζητήσουμε, να μάθουμε για σημαντικές υποθέσεις που έχουν να κάνουν με την ισότητα ανδρών και γυναικών. Δίνω το λόγο λοιπόν στους συναδέλφους. Η κυρία Λεγκρίπ πρώτα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε το χαρτοφυλάκιο για το οποίο είσαστε υποψήφια περιλαμβάνει τα θέματα των καταναλωτών, της δικαιοσύνης αλλά και της ισότητας των φίλων. Η πρώτη φορά που ένα χαρτοφυλάκιο εστιάζει τόσο συγκεκριμένα στα θέματα της ισότητας ανδρών και γυναικών. Αυτό είναι μια βασική αξία, μια θεμελιώδης αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια ιδρυτική ακόμα αξία. Το ερώτημά μου έχει να κάνει με το σχέδιο οδηγίας που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Είπατε ότι εσείς θέλετε να προωθήσετε αυτό το θέμα. Συγκεκριμένα λοιπόν, κύριε Επίτροπε, πώς θα εξασφαλίσετε ότι θα προωθηθεί το θέμα αυτό και ιδίως σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο, γιατί εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη ισορροπία σε αυτό το νομοθέτημα και θα ήθελα να ξέρω τι θα κάνετε έναντι του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γκρίπ για το Για την πρόταση Women on Board συγκεκριμένα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δείξει μια θετική αντιμετώπιση και γι' αυτό το ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη που έχει δείξει. Υπάρχουν πολλές φήμες που κυκλοφορούν γύρω από αυτή την πρόταση υπήρξε μια θύελα μυθοπλασιών και φημών από τα μέσα ενημέρωσης ότι η Κομισιόν θέλει να επιβάλλει στις επιχειρήσεις τον αριθμό γυναικών που θα πρέπει να είναι στα διοικητικά συμβούλια. Ξέρω ότι αυτό θα οδηγούσε σε αντιδράσεις όταν διάβασα όμω την πρόταση, είδα ότι αυτή η πρόταση δεν είναι μονάχα αποτελεσματική, αλλά και απαραίτητη, γιατί θα δώσει περισσότερες ευκαιρίες στις γυναίκες να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια και υπάρχει και η δυνατότητα να εφαρμοστεί με σωστό τρόπο αυτή η πρόταση. Γι' αυτό εγώ θα προχωρήσω σε διαπραγματεύσει και πάλι με το Συμβούλιο για την πρόταση αυτή και θα επανεξετάσω την αποτελεσματικότητα και την εφαρμοσιμότητα αυτή της πρόταση στην πράξη. Είναι σαφής ο στόχος της πρότασης αυτής. Αν είναι 60% των ε, αποφύτων πανεπιστημίων που είναι γυναίκες και έχουν πάρει με μεγάλη επιτυχία το πτυχίο τους. Γιατί δεν βρίσκονται σε υψηλές θέσεις σε όπου το ποσοστό είναι πολύ χαμηλότερο. Και σε ό,τι αφορά την ε, συμμετοχή του σε διοικητικά συμβούλια είναι πραγματικά ζωφερή η κατάσταση. Αυτό είναι λοιπόν ένα θέμα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Θα ξεκινήσω και πάλι τη συζήτηση για το θέμα αυτό με τα κράτη-μέλη και θα προσπαθήσω να υπερκεράσω την ανασχετική μειοψηφία και να εξηγήσω στα κράτη-μέλη ότι είναι πράγματι χρήσιμη αυτή η πρόταση. θα προσπαθήσω να τα μεταπίσω τα κράτη-μέλη. Μπορώ να επανέλθω αργότερα επειδή τέλειωσε ο χρόνος μου. <clears throat> Ευχαριστώ ο κύριος Λάιχτφριντ από τους σοσιαλιστές έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εδώ είμαι, ο μόνος άνδρας σε αυτόν τον κατάλογο από την Επιτροπή Γυναικών. Θέλω ευχαριστήσω τη συναδελφό μου που έθιξε το θέμα των Women on Board, γιατί και το δικό μου ερώτημα περιστρέφεται γύρω από το θέμα αυτό. Ίσως μπορείτε να πείτε πιο συγκεκριμένα τι χρονοδιάγραμμα έχετε για αυτή την νομοθετική πρόταση τι πιστεύετε για τις διαφορετικές θέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν, για τις εξαιρέσεις, για τις κυρώσεις. Ποια είναι τα σχέδιά σας, αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα αφορά την οδηγία για τη μητρική άδεια. Αναφέρατε στις γραπτές σας απαντήσεις ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό γιατί καλύπτει όχι μόνο τις μητέρες αλλά και τους πατέρες τι θα κάνετε λοιπόν για να διατηρήσετε αυτή την οδηγία, τι μέτρα θα λάβετε για να προωθήσετε το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει η κυρία Ούροβα. Σας ευχαριστώ για το θέμα του χρονοδιαγράμματος. Θα ήθελα να εγκριθεί μέσα στον επόμενο χρόνο αυτό το νομοθέτημα. Δεν μπορώ τώρα να είμαι πιο συγκεκριμένη σε σχέση με συγκεκριμένες ημερομηνίες. Αλλά το, η δική μου προσπάθεια θα είναι αυτή και είναι καθήκον μου ενώπιον και του κύριου Γιούγκερ να διευκρινιστεί καλύτερα η κατάσταση με τα κράτη-μέλη. Για την επιβολή κυρώσεων τώρα. Η επιλογή κυρώσεων έχει να κάνει με την αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει με τη διακριτική ευχέρεια που τα χαρακτηρίζει να αποφασίσουν ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να επιβληθούν. Τα κρατημέλη έχουν λοιπόν ένα μεγάλο βαθμό ευελιξίες για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτή την οδηγία και τους κανόνες που συνάπτονται με αυτήν. Εδώ υπάρχει πάντως μια σαφής πρόνοια που αναφέρει ότι τα, τα κύρια κριτήρια θα πρέπει να είναι τα προσόντα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Και εάν υπάρχει, υπάρχουν ίσα προσόντα, η υποστήριξη και η προτεραιότητα θα, θα δοθεί στην ομάδα που υποεκπροσωπείται. Είναι σημαντικό να εξετάσετε λοιπόν την πρόταση και να δείτε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Η γονική άδεια. Για το θέμα αυτό και πάλι πιστεύω θα πρέπει να επανέλθουμε, να ανοίξει και πάλι το ζήτημα αυτό. και φυσικά δεν αφορά μονάχα την άδεια την μητρική αλλά και την πατρική άδεια, η γονική άδεια πρέπει να είναι άδεια αμοιβόμενη για την φροντίδα των παιδιών τους. Θα πρέπει λοιπόν να είναι ενιαίοι οι κανόνες σε σχέση με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την ομάδα των συντηρητικών, η κυρία Φων Στόρκ. Αγαπητή κυρία ε, Γεωρούροβα, είμαι εδώ. Αναφερθήκατε στο θέμα της ε, ίσης αντιμετώπισης ανδρών και γυναικών και της ισότητας των φύλων και το mainstreaming των θεμάτων του φίλου. Το φύλο όμως είναι μονάχα θέμα σεξουαλικό, η διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Γιατί η λέξη φύλλο, με τη σεξουαλική έννοια, έχει αντικατασταθεί με το φύλλο σε μια πιο ουδέτερη ε, έννοια. Μήπως υποκρύπτεται πίσω από αυτό μια πολυμορφία φύλων και αυτό είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά ε, την χάνει διακρίσεων. Το γερμανικό Facebook έχει 16 κατηγορίες και φαίνεται ότι αυτό, αυτές οι βασικές κατηγορίες άνθρας και γυναίκα δεν φτάνουν. Είναι λοιπόν θέμα του τι αισθένεται κανείς. Το φύλλο αυτό είναι το πώς αισθάνεται ο καθένας. Συμφωνείτε με μια τέτοια αντιμετώπιση. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Γιώργο. Εγώ κάπως με από τον αριθμό των φίλων που υπάρχουν στη Γερμανία. Δεν φανταζόμουν ότι μπορούν να είναι τόσα πολλά. Ποια είναι η δική μου λοιπόν αντιμετώπιση για την έννοια του φύλου. Δεν θα προσπαθήσω να αναλύσω από γλωσσική μορφή αυτή τη λέξη. Γιατί δεν θα μπορεί να μην τα καταλήξω σε καλό αποτέλεσμα. Αλλά για μένα η ισότητα των φύλων σημαίνει ότι ο ρόλος των ανδρών και των γυναικών που προκύπτει από τη φυσιολογία τους, από τις κοινωνικές και ιστορικές παραδόσεις. Ξέρω ότι αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία, αλλά για μένα τα θέματα του φύλου σημαίνουν την εξασφάλιση της ισότητας ευκαιριών σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην παιδεία, σε ό,τι αφορά την εργασιακή αγορά, σε ό,τι αφορά θέσεις ε, ευθύνης. Ίσες ευκαιρίες λοιπόν για την πρόσβαση σε υπηρεσίες όλα αυτά λοιπόν τα οποία έχουν στη διάθεσή τους οι άνδρες να είναι διαθέσιμα και στις γυναίκες. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν και δεν νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε γιατί βασίζονται στις παραδόσεις μας. Αλλά θα πρέπει να είμαστε σε θέση να, να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μια γυναίκα πρέπει να έχει αυτό το χάσμα αποδοχών έναντι ενός άνδρα όταν ασκεί την ίδια ακριβώς εργασία με έναν άνδρα ίσον προσόντων. Και εγώ προσωπικά έχω έρθει αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου όχι μονάχα ήμουνα λιγότερο καλά πληρωμένη, αλλά δεν λαμβανόταν υπόψη γνώμη, επειδή ήμουνα γυναίκα και αναφέρομαι στην, στα υπουργικά μου αξιώματα. Πολλές φορές λοιπόν ήμουν σε υποδέστερη θέση λόγω του φίλου μου και αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα αλλάξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτρια, παρακαλώ, κυρία Μπέρντα. Ευχαριστώ πολύ ε, έχετε φτάσει πια στο τέλος μιας ε, μακράς αλλά και περίπλοκης ε, συνεδρίας. Συγχαρητήρια για την αντοχή σας ή μη τι άλλο. στην, προκαταβολική σας, στην προκαταρκτική σας παρέμβαση είπατε ότι θα αγωνιστείτε κατά της βίας. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πώς βλέπετε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση κοινή για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, ευπρόσδεκτη για όλους μας, αλλά συγκεκριμένα θέλω πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια τέτοια προσέγγιση και πρακτικά πώς θα μπορούσατε να εξασφαλίσετε το συντονισμό μεταξύ των διαφορών γενικών διευθύνσεων για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση τη βία της βάρο των γυναικών και ιδιαίτερα θα ήθελα να ρωτήσω πώ σκοπεύετε να συνεργαστείτε με την DG ε, Home για να αναπτύξετε μια ευρωπαϊκή στρατηγική με στόχο την εκρίζωση των ε, του φαινομένου το, του εμπορίου εις βάρος γυναικών, ε, εμπορίου ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ. Η βία εις βάρος των γυναικών πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάθε διαθέσιμο μέσο και σε κάθε ήπειρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι η οντότητα εκείνη η οποία θα εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα κάνει να διαδοθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και έξω από αυτήν, ιδιαίτερα σε χώρες όπου είναι διαδεδομένη ή γενικευμένη καλύτερα πρακτική η βίας βάρος των γυναικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πιστεύω τώρα την ευκαιρία να προσχωρήσει στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που υπογράφηκε τον Ιούνιο και με χαρά διαπιστώνω ότι πολλά κράτη-μέλη, 22 συγκεκριμένα, έχουν υπογράψει την ε, σύμβαση αυτή, 8 εκ των οποίων την έχουν και κυρώσει. Εγώ θα καλούσα όλα τα κρατη να προχωρήσουν στην υπογραφή της ε, συμβάσεως, ώστε να προχωρήσει ιδιαίτερα το θέμα αυτό. Ξέρω ότι σε ένα βαθμό καλύπτονται οι διατάξεις από, την οδηγία της σχετική με τα θύματα ε, βίας. Ε, ξέρω ότι η Ισπανία έχει παραδείγματι ειδική νομοθεσία. Νομοθεσία η οποία ασχολείται ιδιαίτερος με το θέμα της βίας εις βάρος των γυναικών. Και αλλού υπάρχει τέτοια νομοθεσία. Όμως δεν πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο στην νομοθέτηση κειμένων. Πρέπει η κοινωνία ολόκληρη να αντισταθεί και να αντιδράσει. Δεν πρέπει να δεχόμαστε τη βία εις βάρος των γυναικών. Σε είναι κάτι το φυσιολογικό. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους της ε, Γκουε, η επόμενη μιλήτρια. Πράγματι το 2015 θα πρέπει να προχωρήσει στη νομοθετική ρύθμιση για τα θέματα της ισότητας ανδρών γυναικών. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές, έλλειψη γυναικών σε θέσεις ευθύνης, διαφορές μισθολογικές και άλλες μορφές διακρίσεων, όλα αυτά φαίνονται και από τα προγράμματα για την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει επίσης και για τη βία εις βάρος των γυναικών στην πολιτική σφαίρα, λέει η ομιλήτρια. Πώς βλέπετε εσείς πιστεύετε ότι η νέα στρατηγική θα μας δώσει μια σταθερή βάση για τον σεβασμό ε, των δικαιωμάτων των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών για την ανεξαρτητοποίησή τους σε οικονομικό επίπεδο και τι στρατηγικές θα πρέπει να ξεκινήσουμε έτσι ώστε να ενισχύσουμε το νομικό πλαίσιο προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ισότητας των ευκαιριών. Ε, θα πρέπει η χρηματοδότηση για τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι πιο ικανοποιητική από τη σήμερα στις διάφορες χώρες. Σας ευχαριστώ. Εφόσον με επιβεβαιώσετε σαν επίτροπο για τα θέματα της ισότητας των φύλων, θα αναλάβω η υπηρεσία τη στιγμή ακριβώς της διατύπωσης της τελικής στρατηγικής για την ισότητα των ευκαιριών και της επίλυσης των προβλημάτων των γυναικών στην κοινωνία. Η νέα αυτή στρατηγική θα πρέπει να βασίζεται όμως σε συγκεκριμένα στοιχεία και δεδομένα τα οποία να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα θα πρέπει να βασίζεται σε μια στενή εταιρική σχέση με όλους αυτούς που μπορούν να επηρεάσουν θετικά την κατάσταση των γυναικών. Είτε είναι οι κρατικές οργανώσεις, είτε είναι επαγγελματικέ οργανώσεις. Έχω την αίσθηση ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης και ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο να βασίζεται σε μελλοντικές νομοθετικές και μη νομοθετικές λήψεις μέτρων. Δεν θέλω να τα απαριθμίσω όλα αυτά τώρα. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να είναι καρπός μια συζήτηση που θα γίνει και σε επίπεδο επιτροπής. Η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης έχει αρκετούς πόρους για την στήριξη ορισμένων προγραμμάτων και μία από τις αρμοδιότητες μου θα είναι να διασφαλίσω τη σωστή χρήση αυτών των πιστώσεων. Και θα πρέπει επίσης να πάρουμε και αποφάσεις ε, σχετικά με την ανάγκη ή μη της δημιουργίας μιας ενδιάμεσης έκθεσης, αξιολόγησης. Γιατί όπως είπα η στρατηγική αυτή θα πρέπει να υπευθυμενοποιεί όλους όσους συμμετέχουν στις διαδικασίες. Για την ομάδα των Πρασίνων, η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχουμε αναφερθεί, λέει η κυρία Ρέντ, και για την πρόταση Women on Board, ε, σε υπεύθυνε θέσεις γυναίκες. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μένει να γίνουν προς την κατεύθυνση αυτή. Πώς αυτές τις αρχές ε, τις οποίες ε, θέλουμε να εφαρμόσουμε θα πετύχουμε να τις εφαρμόσουμε. Και τι γίνεται με την ισότιμη εκπροσώπηση ανδρών γυναικών τουλάχιστον στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για, τις, για τα κράτη-μέλη να προτείνουν γυναίκες για την συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα στραφείτε στα κράτη-μέλη πριν από τις επόμενες εκλογές έτσι ώστε να προτείνουν έναν άνδρα και μία γυναίκα υποψηφίους έτσι ώστε να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στα φύλλα και αν υπάρχει μια θα έλεγα διάκριση σε σχέση με, με τον ορισμό ε, του φίλου υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο της Judith Butler η οποία ε, θα σας ενημερώσει σωστά για το τι σημαίνει το φίλο του ανθρώπου. Ευχαριστώ κυρία Ρένκε. Νομίζω ότι πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δίδει το σωστό παράδειγμα. Και εγώ ε, όταν είδα το ποσοστό 9 γυναίκες ε, στους 28 νομίζω, δεν θυμάμαι ακριβώς, είναι κάτι το οποίο δεν είναι ε, κάτι το οποίο με ικανοποιεί και φυσικά δεν είναι κάτι το οποίο σέβεται τις προτάσεις τις οποίες περιλαμβάνει η οδηγία Women on Board, γυναίκες σε θέσεις ευθύνη. Και δεν ξέρω ακριβώς τώρα πώς θα καλυφθούν οι διάφορες θέσεις στις γενικές διευθύνσεις, αλλά νομίζω ότι και εκεί το ποσοστό των γυναικών είναι ιδιαίτερος χαμηλό. Λοιπόν, ε, η υποχρέωση την οποία καλούμε συνεπώς να αναλάβω και το κάνω αυτό, είναι να παρουσιάσω προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αύξηση της αντιπροσωπευτικότητας της, ε, του αριθμού των γυναικών σε υπεύθυνε θέσεις. Σχετικά τώρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επόμενη, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ εγώ να επηρεάσω, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να προτείνω την αύξηση του αριθμού των γυναικών και σας ευχαριστώ και για τη σύσταση του βιβλίου της Μπάτλερ. Ευχαριστώ. Η κυρία Αιούτο από το FND. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, επιθυμητή είπατε ότι είναι η ομοιογένεια ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα για τις νέες μητέρες. Ε, τα προβλήματα που δημιουργούνται στην αγορά εργασίας μετά τη γέννηση του παιδιού είναι κάτι το οποίο χειροτερεύει την κατάσταση των ε, νέων γυναικών. Ε, το τι θα κάνουν οι γυναίκες με τα παιδιά είναι μια ανησυχία η οποία επηρεάζει την είσοδο των γυναικών στις αγορές, στην αγορά εργασίας. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να βοηθήσει τις χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει αρκετά να καλύψουν την ανησυχία αυτή. Πολλές φορές ε, οι υπηρεσίες ε, για τα παιδιά ε, δεν είναι ικανοποιητικές από πλευράς κρατικής και συνεπώς αναγκάζονται οι νέοι γονείς να στρέφονται σε εναλλακτικέ δομές φροντίδας των παιδιών οι οποίες είναι ιδιαίτερα υψηλού κόστους. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Ήδη πριν ξεκινήσει η κρίση ήταν σαφές ότι υπάρχει άλλωστε ένας όρος στην κοινωνιολογία ο οποίος λέγεται η αύξηση των γυναικείων χαρακτηριστικών της ένδυας. Αυτό, ε, η ορολογία αυτή αποδεικνύεται από τους αριθμούς οι οποίοι δείχνουν ότι οι συνθήκες με τους οποίους βιώνουν οι γυναίκες έχουν χειροτερεύσει και αυτό κυρίως αφορά τις νέες μητέρες. Αναφερθήκαμε σε προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε τομείς όπως η, μητρική άδεια και για την στήριξη που θα πρέπει να δοθεί στη μητέρα ή στον πατέρα κτλ. Το θέμα δεν είναι απλά ε, η στήριξη προς ένα πρόσωπο, προς ένα γονέα. Το θέμα είναι να μπορέσει η γυναίκα να ξεφύγει από την ε, πολλαπλή πίεση την οποία, ε, την εφίσταται για να φροντίσει σωστά τα παιδιά της και πολλές φορές να φροντίσει σωστά και τους γονείς της. Και αυτό είναι δυστυχώς ένα νέο φαινόμενο. Είναι γυναίκες οι οποίες ε, έχουν θέσεις εργασίας αλλά δεν μπορούν να τις καλύψουν ικανοποιητικά και συνέπεια είναι να έχουν οικονομικά προβλήματα γιατί έχουν πάρα πολλή δουλειά στο σπίτι. Υπάρχει μια δυνατότητα λύσης ε, να χρησιμοποιηθούν τα διαφθορτικά ταμεία, ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι κάτι με το οποίο έχω απασχοληθεί στο παρελθόν. Υπάρχουν εκεί πιστώσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται μόνο για την καταπολέμηση της φτώχειας αλλά και για την εναρμόνιση ή μάλλον καλύτερα τον αρμονικό συνδυασμό της οικογενειακής από τη μία ζωής και της επαγγελματικής δραστηριότητας από την άλλη πάρα πολύ σωστά είπατε ότι τα προβλήματα δεν είναι τα ίδια βέβαια όλα σε κράτη-μέλη, γι' αυτό ας δούμε αναλογικά πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ευχαριστώ. Η κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, ως νομομαθής, συμφωνείτε μαζί μου για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Συμφωνείτε μαζί μου ότι πρέπει να υπάρξει προστασία αυτών των δικαιωμάτων. Και επίσης αυτό πάλι είναι θέμα ίσων ευκαιριών. Υπάρχουν διαφορετικά είδη παραβιάσεων των δικαιωμάτων των εργαζομένων που έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο στις γυναίκες γιατί έχουν και οικογενειακές ευθύνες συγχρόνως. Σκέφτομαι το χρόνο εργασίας, τη δυνατότητα άδεια και την αδυναμία του να μπορούν να προγραμματίσουν το πότε θα πάρουν άδεια, τον κίνδυνο να χάσουν τη θέση εργασίας τους, το φόβο να χάσουν την εργασία τους, το... Όλα αυτά λοιπόν προσδιορίζουν τη ζωή αυτών των γυναικών. Τι θα κάνετε λοιπόν σε σχέση με τα φαινόμενα αυτά τα οποία αφορούν εκατομμύρια γυναίκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω στα κράτη, τα νέα κρατημέλια όπω στη χώρα μου την Ουγγαρία. Ε, ναι. Υπάρχουν δικαιώματα εργοδοτών και εργαζομένων και προσπάθειες που αναπτύσσονται από όλα τα κράτη-μέλη. Και έχω συμμετάσχει σε αρκετές τριμερείς συζητήσεις, ώστε να γνωρίζω ότι πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των εργοδοτών και αυτών των εργαζομένων. Εγώ ως δικηγόρος λοιπόν θα απαντήσω καταφατικά στην ερώτησή σας. Τα πάντα θα κρυθούν από την ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών των, ε, συμφερόντων των δύο αυτών ομάδων. Και ο εργαζόμενος να έχει τα δικαιώματά του, αλλά και ο εργοδότης να μπορεί να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας για να τις ε, ε, αξιοποιήσουν, για να μπορούν να δουλεύουν εκεί οι εργαζόμενοι. για τις συνέπειες για τη ζωή της γυναίκας, ε, το άγχος, την αδυναμία να πάρει άδεια και την πίεση που συνεπάγονται όλα αυτά. Είναι φαινόμενα και της σύγχρονης κοινωνίας. Είναι πολλές οι πιέσεις που υφίστανται οι γυναίκες, πολλές οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω μπορεί να αναπτύξει εκστρατείες για ευαισθητοποίηση αλλά και να υιοθετήσει νομοθετικά ε, κείμενα. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε το κοινωνικό ταμείο γιατί υπάρχουν κονδύλια ειδικά για τον τομέα αυτών και για την Ουγγαρία που θα βοηθήσουν στη βελτίωση της κατάστασης. Πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα τώρα στην ε, Τσεχική Δημοκρατία. Θέλουμε να αξιοποιείται περισσότερο, πιο συχνά, η μερική επασχόληση για ε, ομάδες ανθρώπων που θα μπορούσαν να αναλαμβάνουν τα παιδιά σε προσχολική ηλικία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κοράτσα Πίλτ, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ, κυρία Ρόβα. Ελπίζω να αντέξετε να τα βγάλετε πέρα και με τις τελευταίες δύο ερωτήσεις. Μία στις τέσσερις γυναίκες στην Ευρώπη σήμερα εφίσταται σωματική βία, ε, μία στις ναι. δέκα σεξουαλική, γενετήσια βία, εκμετάλλευση, βία εις βάρος των γυναικών. Ε, αναφερθήκατε και εσείς στην ε, κλειτοριδεκτομή και σε άλλα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ που τα αναφέρατε αυτά. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω πώς μπορείτε να ε, σταθείτε ε, στο ύψος σας ενώπιον των κρατών μελών για να αντιμετωπίσουν τα θέματα της ε, μετάλλευσης των γυναικών, των παιδιών, των θυμάτων, των εγκλημάτων αυτών και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μικρά κορίτσια. Δεύτερον, είπατε ότι θα πρέπει η Επιτροπή να κυρώσει την Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, της Κωνσταντινούπολης, όπως λέγεται, για την προστασία των γυναικών και γιατί μόνο οκτώ κράτη-μέλη έχουν κυρώσει μέχρι στιγμής. Θα αναλάβετε πρωτοβουλία για να πιέσετε τα κράτη-μέλη για να προχωρήσουν σε τοχετερή κύρωση όσο δεν το έχουν πράξει και πώς θα γίνει η κύρωση πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης δεν θέλω να ρωτήσω αν έχετε μια στρατηγική για την εκρίζωση και πρόληψη στη βία ε, εις βάρος των γυναικών. Ε, και όταν λέω στρατηγική εννοώ τι είδους συγκεκριμένες δράσεις μπορείτε να μας υποβάλλετε. Απάντηση. Όπως είπα και νωρίτερα θα μεριμνήσω να κυρωθεί η σύμβαση από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αποτελεί, πιστεύω, ένα σημαντικό βήμα πρόοδου, όχι μόνο ως προς το σεβασμό των κανόνων, αλλά και ως προς την ευαισθητοποίηση του κοινού, να αντιληφθεί δηλαδή ο καθένας ότι δεν είναι φυσιολογικό το να, να υφίστανται βία, είτε γυναίκες είτε νεαρά κορίτσια. Ε, είναι αδύνατο να εκρίζωθεί πλήρως το φαινόμενο αυτό δυστυχώς στην κοινωνία. Αλλά πρέπει να αξιοποιήσουμε κάθε νομοθετικό και μη νομοθετικό μέσο. Η κύρωση της συνθήκης ήταν το πρώτο βήμα το οποίο θα ήθελα να προωθήσω. Και θα ήθελα να πιέσω τα κράτη-μέλη να κυρώσουν τη σύμβαση στη διάρκεια του επόμενου έτους θα ήθελα να οργανώσω μια σειρά από ε, διαλόγους, συζητήσεις, δημόσιες για το θέμα της βίας εις βάρος των γυναικών, από τις οποίες θα περίμενα να προκύψει απάντηση για το αν χρειάζεται ειδική νομοθεσία όπως υπάρχει στις ΗΠΑ. Θα είναι και αυτό λοιπόν ένα κομμάτι της δουλειάς μου με μια, μέσα σε μια γενική στρατηγική. Θα είναι μια απάντηση στο ερώτημα του τι νομοθετικά βήματα χρειάζονται. Κάτι ακόμα ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό νομίζω, το πώς τα ίδια τα κράτη-μέλη βλέπουν, τι είδους θεώρηση έχουν τα κράτη-μέλη για το πρόβλημα της βίας των γυναικών. Και αν το την χαρακτηρίζουν ως έγκλημα, ως αδίκημα. Πρέπει να κοιτάξουμε δηλαδή αν προβλέπονται αυστηρότερες ποινές σε περίπτωση της άσκησης βίας εις βάρος των γυναικών σε σχέση με την ε, κοινή βία. Και όταν ε, και θα πρέπει να κοιτάξουμε αν υπάρχουν προληπτικά μέτρα για την αποτροπή της βίας βάρος των γυναικών στα κράτη-μέλη. Τελευταία ομιλήτρια από την ομάδα των Σοσιαστών, κυρία Αρένα. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να κλείσω αυτή την ε, μακρά σειρά ερωτήσεων. Θέλω να σταθώ σε ένα ερώτημα που έχει να κάνει με τη, τη μητρική άδεια. Είπατε ότι υποστηρίζετε μια συζήτηση για την ε, άδεια αυτή. Το ερώτημα μου είναι πιο συγκεκριμένα. Σήμερα υπάρχει ένα κείμενο το οποίο θα σας επέτρεπε να προχωρήσετε αρκετά γρήγορα και το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι διαπραγματεύσεων του Συμβουλίου και θέλω να ξέρω αν θα λειτουργήσετε από τη βάση αυτού του κειμένου που θα σας επιτρέψει να πάτε πολύ πιο γρήγορα και το οποίο είναι ο καρπός της εργασίας και της επεξεργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια θα είναι η θέση του Συμβουλίου, αλλά νομίζω ότι εμείς θεωρούμε πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό το έγγραφο ως βάση. Δεύτερον, στην απάντησή σας για τα γραπτά, στα γραπτά ερωτήματα είπατε ότι η προηγούμενη στρατηγική είχε οδηγήσει σε ορισμένα αποτελέσματα για τη στρατηγική υπέρ των τη ισότητα ανδρών και γυναικών, αλλά υπάρχει πολλοί δρόμος να διατρέξουμε και αναφέρατε τα χάσματα σε σχέση με την, τις και τις συντάξεις, τη βία, την ένδια των γυναικών. Τι θα κάνετε συγκεκριμένα για να υπάρχει μια πραγματικά αποτελεσματική στρατηγική μετά το 2015 και πώς θα πείσετε όλους του συναδέλφους σας στην Κομισιόν για την ενσωμάτωση της διάστασης του φίλου σε όλες τις πολιτικές γιατί αφορά όλους τους επιτρόπους που βρίσκονται σε ακροάσεις και οι οποίοι μερικοί από αυτούς έχουν δυσκολία με την ισότητα των φίλων από ό,τι ξέρω. η σαφής μου απάντηση είναι ναι σε αυτά τα ερωτήματα. Πράγματι θέλω να συνεχίσω να εργάζομαι για επί των προτάσεων που είναι τώρα στο Συμβούλιο, στη συζήτηση του Συμβουλίου. Θα το συζητήσω και με την κυρία Τάισεν, γιατί αφορά και τα θέματα της απασχόλησης. Και θέλω να αντιμετωπίσω τα διαδικαστικά προσκόμματα γιατί έχει εμποδιστεί για πολύ χρονικό διάστημα η επεξεργασία αυτής της προτάσεως και πρέπει να ανοίξει και πάλι η επεξεργασία της. Για τη στρατηγική που αναφέρατε και πώς θα εξασφαλίσουμε ότι αυτή η στρατηγική μπορεί να είναι αποτελεσματική. Χωρίς ειδικέ προτάσεις, τι μπορούμε να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε ισότητα απασχόληση, αντιμετώπιση της ένδυας, της βίας που στρέφεται ειδικά κατά των γυναικών, της καλύτερης πρόσφασης στην παιδεία και την υγειονομική περίθαλψη και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία δεν μπορείτε να τα απαριθμίσω χωρίς να είμαστε συγκεκριμένοι για τα θέματα αυτά, χωρίς να έχουμε συγκεκριμένες λύσεις και χρονοδιαγράμματα, δεν μπορεί να λειτουργήσει καμία στρατηγική. Αυτό το οποίο μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι δεν θα προετοιμάσω κάποια στρατηγική μόνο για να είναι στρατηγικές, οι οποίες στη συνέχεια θα τεθούν στον κάλαθο των αχρήστων ή σε κάποιο ράφι. Θέλω αυτές οι στρατηγικές να είναι αποτελεσματικές. Δεν θέλω